Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα στη σημερινή συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι 3 και 8, πρέπει να ξεκινήσουμε Σημείο που ένα έγκριση ημερησία διάταξη. Έχετε σχόλια. Δεν έχετε σχόλια. Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη επομένω. Σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της 29ης Νοεμβρίου 2016 ελήψη σχολείων μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Τέσσερα. Ανταλλαγές απόψεων με τον κύριο Μπέργκε Μπρέντε, τον Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, εξ ονόματος όλου μας, να Καλωσορίζω τον κύριο Μπέγκε Μπρέντε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι ο Υπουργό Εξωτερικών τη Νορβηγία, όπω ξέρετε, και τον συνοδεύει η Νορβηγή ε, πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία επίση καλωσορίζω. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία σα, κύριε Μπρέντε, να απευθυνθείτε ενώπιον τη Επιτροπής μα και να μα παρουσιάσετε την Νορβηγική θέση για διάφορα διεθνή θέματα, ιδίως με εστίαση στην περιοχή της Αρκτικής και εν ώψη της χθεσινής, ε, της μάλλον τη αυριανής ψηφοφορίας τη κοινή έκθεση Envy Affet για την περιοχή της Αρκτικής. Η Νορβηγία βέβαια δεν είναι μέρος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένας στενός φίλος, σύμμαχος και εταίρος για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένα αξιόπιστο σύμμαχος και εταίρο έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ στενέ οι σχέσει μα με την Νορβηγία. Πριν από τη σημερινή συνεδρίαση συναντηθήκαμε με τον κύριο Μπρέντε και συμφωνήσαμε ότι θα λάβει το λόγο για 15 περίπου λεπτά και μετά θα είχαμε την ευκαιρία να <clears throat> θέσουμε ερωτήματα κάνουμε σχόλια και μετά θα συνοψίσει ώστε το πρώτο αυτό θέμα να μπορέσει να περατωθεί μέχρι τις 4. Σε ό,τι αφορά τις στενές σχέσεις της Νορβηγίας με την κοινή αγορά, την συνεργασία μας για αποστολές της ΚΕΠΑ, για πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, όπως η προσπάθεια συμφιλίωσης Ισραήλ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και θα θέλαμε να ακούσουμε την απόψή σας κύριε Μπρέντε και στο δεύτερο τμήμα. Εάν θέλετε θα μπορούσατε να μπείτε και σε περισσότερα λεπτομέρεια για τα θέματα της ακτικής, για τις στρατηγικές προτεραιότητες της ε, Νορβηγίας που είναι οι περιοχές κοντά στον Ακτικό Κύκλο και μέσα στον Ακτικό Κύκλο. Έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Μπρέντε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάλιστε και σας ε, συγχαίρω για την νέα αυτή σας ε, θέση ως ε, πρόεδρος αυτής της πολύ σημαντικής επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου προσφέρεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους τους βουλευτές σε αυτή την επιτροπή. Επίσης, ο πρόεδρος ανέφερε εμφατικά ότι πράγματι αισθανόμαστε ότι είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι. Νομίζω ότι η συνεργασία μέσω της κοινή αγοράς βεβαίως και είναι ένα στοιχείο που μας καθιστά στενούς συμμάχους, αλλά πέρα από αυτό, στη σημερινή εποχή, θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω και εγώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά κοινή αγορά, η εσωτερική αγορά, είναι κάτι παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δομή επί της οποίας συμφωνήσαμε όλοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η ΕΚΑΧ, η οποία εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το προπύργιό μας ε, κατά του προστατευτισμού, του εθνικισμού και επίσης και του λαϊκισμού. Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η εγγύηση για την Ευρώπη, μια Ευρώπη όπου θα παραμείνει μια περιοχή με κράτος δικαίου. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι σε αυτό το κομμάτι του κόσμου δεν θέλουμε να πάρουμε αυτά που είναι στο παρελθόν και να τα μεταφέρουμε στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο για μένα η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και γι' αυτόν επίσης το λόγο εγώ επιθυμώ να έχω μία παλόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που ε, θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ε, προκλήσεις. όπως είπε και ο Τσότσιλ, προς τα πίσω μπορεί κανείς να κοιτάει προς τα μπροστά, μάλλον να παρατηρεί προς τα μπροστά, απλά να κοιτάει. Σήμερα η Ευρώπη είναι πιο εύθραυστη. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πιο αδύναμη η Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές ε, προκλήσεις ε, που πλήττουν την Ευρώπη και εσείς ως μέλη της Επιτροπής αλλά και εσείς ε, πρόεδρε πιστεύω ότι αισθάνεστε αυτά σε καθημερινή βάση. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Αναφέρομαι προφανώς σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η γεωγραφική απόσταση δεν σημαίνει πια ότι είμαστε μακριά από τα προβλήματα. Τις τελευταίες ημέρες ε, διεπιστώνουμε ότι η εξωτερική πολιτική έχει γίνει πλέον και εσωτερική πολιτική. Έχει γίνει μια πραγματικότητα ε, στην καθημερινότητα των χωρών. Άρα δηλαδή αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα και πρέπει να ε, συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα κόσμο με λύσεις που ωφελούν όλους. Εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο δραματίζει σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης. Και όπως σας είπα, πραγματικά χρειαζόμαστε το να αναλαμβάνουν ε, όλοι περισσότερες ε, ευθύνες όσον αφορά την ασφάλεια των κρατών. Αυτό είναι καθοριστική σημασία, άρα στον τομέα αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Μπορείτε να βασιστείτε στη Νορβηγία. Εμείς παραμένουμε απόλυτα προσιλωμένοι στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και δεν είμαστε μέλλον, αλλά είμαστε πολύ στενά συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα του, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Και εγώ πιστεύω ότι ως κράτος ε, συμβάλλουμε και εμείς ε, το δικό μας, ε, αυτό που μας αναλογεί. Μέχρι το 2021 η Νορβηγία θα προσφέρει, θα συνδράμει 2,8 δις ευρώ για να στηριχθούν 15 κράτη-μέλη μέσα από δικ κάμα σε κονδύλια για να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική. Βέβαια κύριε Πρόεδρε υπάρχει ένα θέμα που μας αποσχολεί όλους, το Brexit. Το Brexit είναι σαφές ότι θα έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας. Και το Brexit εμφανίζεται σε μια περίοδο όπου έχουμε δαπανίσει τα κονδύλια μας για άλλες προκλήσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, η Ρωσία, τα θέματα της μετανάστευσης, οικονομική και κοινωνική μετανάστευση, η κατάσταση στο Μαγκρέπ, στο Σαχέλ έχουμε νέα κυβέρνηση στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε και αυτήν πρέπει κάπως ε, να την αντιμετωπίσουμε και οφείλουμε να βρούμε τους αποτελεσματικούς τρόπους για να κάνουμε όλα αυτά. Και να ξαφνικά έρχεται και το Brexit. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα για όλους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι όσον αφορά τα τεκτενόμενα στις ΗΠΑ δήλωσε ότι επιθυμεί να είναι πλήρως ενημερωμένη ε, και θα δει και πώς θα χειριστεί το θέμα του Brexit. Όπως είπε και ο πρόεδρος, η Αρκτική είναι και αυτή ένα θέμα που αφορά όλους μας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει για την Αρκτική. Η δική μου άποψη είναι ότι ο κόσμος αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά δυστυχώς η Αρκτική αλλάζει ακόμα πιο γρήγορα. Ε, η περιβαλλοντική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής πρέπει να προχωρήσουν μαζί. Μερικοί λένε ότι αυτό μοιάζει λιγάκι με τετραγωνισμό του κύκλου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε μπορέσει να καταδείξουμε ότι η Αρκτική είναι μια περιοχή όπου υπάρχει ε, οικονομική συνεργασία, σταθερότητα, ειρήνη και προβλεψιμότητα. Έχουμε εφαρμόσει όλα τα περιοριστικά μέτρα που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση σε αυτά που συνέβησαν στην Κρυμαία και στον Ντομπάς και παράλληλα μπορέσαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Ρωσία στο Βορρά. Συνεχίσαμε τη συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα, στην πυρηνική ασφάλεια και θα ήθελα να πω ότι κατορθώσαμε τα αποθέματα ψαριών να τα διαχειριστούμε και αυτά αποτελεσματικά. Ένα εκατομμύριο τόνους μπακαλιάρου στον βορρά. Αυτό είναι το ε, ε, απόθεμα ψαριών. Χρησιμοποίησαμε βέβαια για να τα πετύχουμε όλα αυτά και τις ε, συμβουλές των επιστημόνων και των ειδικών. Αυτά τα καταφέραμε από κοινού με τη Ρωσία και ας μην ξεχνάμε ότι ε, το κάναμε, το πετύχαμε, ενώ υπήρχε μεγαλύτερη ένταση από ό,τι κατά το παρελθόν. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική μας για την Αρκτική είναι η Αρκτική να παραμείνει ειρηνική, σταθερή και ένα προβλέψιμο μέρος του κόσμου. Ε, νομίζω ότι Επ' αυτού συμφωνούν ε, και τα κράτη της ε, Αρκτικής, γιατί συμφωνούν ότι ε, ο νόμος της θάλασσας είναι το πλαίσιο. Είναι ένα είδος συντάγματος για την Αρκτική και είναι πάντα ένα καλό πλαίσιο για να ξεκινήσει κανείς τη συνεργασία στις χώρες της Ακτικής ε, έχουμε χώρες ε, σε τρεις υπήρους οι οποίες βρήκαν έναν τρόπο να συνεργάζονται και να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Οι πέντε παράκτες χώρες ε, στον Αρκτικό ωκεανό συμφώνησαν ότι οι επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις στην υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου αυτό είναι τουλάχιστον μια ε, ελπίδα που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο. Είναι αυτονόητο κάτι τέτοιο. Επίσης, ε, Υπάρχει ένα σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από δικές σας ε, συμβουλές βλέπουμε λοιπόν ότι κατά τα επόμενα έτη θα υπάρχει αυξημένη, ε, αυξημένα αιτήματα, θα υπάρχουν για τις ε, πρώτες ύλες της Αρκτικής. Θα αυξηθεί γενικά ο πληθυσμός της γης, άρα ε, οι ποσότητες πρωτεΐνης που θα είναι απαραίτητες θα αυξηθούν και αυτές. Ε, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, ε, όπως σας είπα, θα χρειάζεται περισσότερα τρόφιμα, ενέργεια, ορυκτά, θα πρέπει να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες. Ακόμα και αν κατορθώσουμε να αποσυνδέσουμε την αύξηση του πληθυσμού από την οικονομική ανάπτυξη, παρόλα αυτά πρέπει να δεχτούμε ότι θα υπάρχει αύξηση της ζήτησης. Τη ζήτηση ε, κυρίως σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ζημιά στο περιβάλλον, ε, αυτά πρέπει πάντα να τα έχουμε κατά νου. Η Αρκτική είναι κυρίως ωκεανός και η μπλε οικονομία ενέχει πολλές ελπίδες για νέες επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση. Στη Νορβηγία η χρήση των πρώτων υλών του ωκεανού ε, αποτελεί τη βάση της οικονομίας μας. Και αυτό θέλω να μεταφέρω σε εσά, διότι αν δεν υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι στην Αρκτική, έστω πάρα πολύ λίγοι, 3-4 αυτό είναι ένα θέμα, αλλά ξέρω ότι ο πρόεδρος και εσείς γνωρίζετε η Νορβηγία έχει εκμεταλλευτεί ε, τους, ε, τις πρώτες ύλες εδώ και πάνω από 10.000 χρόνια. Έχουμε 10% του πληθυσμού μας που ζει στον αρκτικό κύκλο. Δεν ισχύει για κανένα άλλο κράτος αυτό. Το 80% των ε, παράκτηων περιοχών μας βρίσκεται βόρεια της Αρκτικής. Περίπου τα 2 τρίτα των εσόδων μας από τις εξαγωγές ε, προέρχονται από δραστηριότητες ε, στη θάλασσα και από θαλάσσιους ε, πόρους. Γι' αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προάγουμε Μας ενδιαφέρει λοιπόν να προάγουμε τη διαχείριση όλων αυτών των πρώτων υλών. Εδώ και δεκαετίες μπορέσαμε να έχουμε κάποια ισορροπία στα οικοσυστήματα και ίσως αυτό να σας φανεί μια σύμπτωση Πριν από 10 χρόνια παρουσίασα την πρώτη λευκή βίβλο Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε αυτή την επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση ε, γιατί εκεί αναφέρεται η εφόρος χρήση των πόρων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και πρέπει να υπογραμμιστεί είναι καταδείξαμε ότι είναι απολύτως ε, εφικτό ε, να συνδυάσουμε την αλληλεία, τις ιδιωτοκαλλιέργειες, την αυτιλία, την ενέργεια και ένα υγιές ε, θαλάσσιο περιβάλλον. Η περιοχή αυτή της Αρκτικής παραμένει ε, ένας ε, πολύ καθαρός, μια πολύ καθαρή περιοχή του κόσμου. Κύριε Πρόεδρε, Ε, κύριε Πρόεδρε, αυτά αφορούν την Αρκτική και αυτά αφορούν και στη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική ασφάλειας. Ε, νομίζω η συνεργασία μας ε, είναι πολύ στενή. Θα έχουμε την επόμενη κοινή συνάντησή μας, ε, την συνάντηση των δωρητών, αρχές Μαΐου για την Παλαιστίνη. Και εκεί είναι η μόνη περίπτωση όπου θα έχουμε στο ίδιο τραπέζι Παλαιστίνιους με Ισραηλινούς. Ε, μπορούμε να ε, λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και να στηριχθούν οι απαραίτητες κρατικές δομές στη Ραμάλα. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με τη Συρία. Η Νορβηγία είναι εκείνη η οποία δρομολόγησε τη συνδιάσκεψη για τη Συρία που έλαβε χώρα πέρυσι το Φεβρουάριο σε συνεργασία με τη Γερμανία, το Κουβέιτ. Ε, ε, τώρα έχει ε, ανακοινωθεί μια περαιτέρω συνάντηση από την κυρία Μογκερίνη. πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία ε, θα κρίνουν κατά πόσον τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό ισχύει για όλους. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε να ε, επεξεργαζόμαστε πολιτικές λύσεις με την έχουμε την υποστήριξη του κύριου Στέφαν Δεμεστούρα σε αυτό το θέμα. Συνεργαζόμαστε για τη Λιβύη, για την Κολομβία. Η Νορβηγία προσπαθεί να διευκολύνει την Κολομβία και βλέπω έχουν εκφραστεί και άλλες απόψεις για το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την Κολομβία. Και τέλος, ως προς τα δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να είμαστε ε, πολύ προσεκτικοί μετά τις τελευταίες εξελίξεις γιατί ενδεχομένως αυτή να είναι η επόμενη πρόκληση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Εμείς σας ευχαριστούμε, ε, κύριε Υπουργέ Μπρέντε, για τα όσα μας είπατε. Προτείνω τώρα να εκφραστούν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ας προσπαθήσουμε να μην ξεπεράσει ο κάθε ομιλητή τα δύο λεπτά, μετά θα έχουμε και άλλες ερωτήσεις ε, και τη δυνατότητα για άλλες παρεμβάσεις. Ε, ο κύριος Γκάλερ από το ΕΛΚ και επίσης ε, και σκιώδης ε, για την έκθεση για την Αρκτική. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Υπουργέ. Εδώ βρίσκομαι, εδώ είμαι. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, ε, αναφορά που κάνατε μεταξύ άλλων και στην Αρκτική. Εγώ και την προηγούμενη θητεία ήμουν εισηγητής ε, για τα θέματα της Αρκτικής και μάλιστα είχαμε και την ευκαιρία ε, να, έχω, να δεχτούμε την φιλοξενία σας στο Όσλο και συζητήσαμε επίσης, περιδιαβήκαμε και με ένα ερευνητικό σκάφος τη περιοχή Αρκτικής και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ε, παλιότερα είσαστε και Υπουργός Περιβάλλοντος και τώρα Υπουργός Εξωτερικών και Πρέπει να πω ότι εγώ πάντα έλεγα και λέγαμε στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένη προσέγγιση ε, όταν μιλάμε για την Αρκτική, δηλαδή μια προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία περιβαλλοντικά, ναυτιλιακά, νομικά κτλ. και δεν αλλάζουμε την. Ε, και φαίνεται ότι τώρα έχει αλλάξει λίγο η προσέγγιση σας ε, και δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο περιβάλλον. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν σα ρωτώ οι συνεργάτες σας ε, έχουν ελέγξει, φαντάζομαι, επανειλημμένα το προσχέδιο της έκθεσής μας και θα θέλαμε να μας πείτε εάν υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια σημεία μάλλον, στα οποία θεωρείτε ότι έχουμε ε, υπερβεί τα των αρμοδιοτήτων μας, εάν υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία ε, ενδεχομένως θα θέλατε να προσέξουμε περισσότερο. Υπάρχουν τρεις χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη του Συμβουλίου της Αρκτικής ε, και επίσης υπάρχουν ε, και ε, δεν έχουμε πλέον παράκτιες χώρες, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα όσον αφορά το θέμα αυτό και εάν έχετε κάποια στοιχεία τα οποία πνέκτης θέλετε να σημειώσετε. Ευχαριστώ πολύ από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, λέει κύριος Φρόγκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για το, την παρουσίασή σας. Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία παρουσιάσατε ήταν μια ροδόχρουση εικόνα των σχέσεων της χώρας σας. Με τη γειτονική Ρωσία ένιωσα και κάποια έκπληξη ακούγοντας αυτά που είπατε. Η δική μου εντύπωση ήταν ε, ότι οι σχέσεις σας με τη Ρωσία είχαν γίνει τόσο αρνητικέ, μάλλον οι σχέσεις της Ρωσίας και τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν γίνει τόσο αρνητικές τον τελευταίο καιρό που δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι θετικό για οποιαδήποτε άλλη χώρα τη περιοχή. Αλλά εκπλήσωμαι και ίσω χαίρομαι που είπατε ότι φαίνεται ότι υπάρχουν σχετικά καλές σχέσεις μεταξύ της Νορβηγίας και της Ρωσίας. Είδατε την σειρά το Occupied, την νορβηγική αυτή σειρά της τηλεόρασης. Όταν τα βλέπω αυτά, ναι, καταλαβαίνετε τι λέω. Νιώθω μεγάλη έκπληξη γιατί αυτή η τηλεοπτική σειρά είχε παρουσιάσει με πολύ πιο ζωφερά χρώματα τις προθέσεις των Ρώσων στην γεωγραφική σας περιοχή και γι' αυτό με εκπλήσει αυτό το οποίο είπατε. Θα ήθελα λοιπόν να πείτε λίγα περισσότερα παρά το γεγονό ότι όλοι φυσικά ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον και οι Ρώσοι όσο και εμεί, για το πώ βλέπετε την ανάπτυξη των σχέσεών σα με τη Ρωσία. Και το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το Brexit. Δεν χρειάζεται να σα το εξηγήσω για το ότι πολλοί έχουν πει ότι η Μεγάλη Βρετανία θέλει να ακολουθήσει το ρόλο της, το παράδειγμα μάλλον της Νορβηγίας σε ό,τι αφορά τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο έχετε κάποιες ιδέες για το κατά πόσο αυτό θα ήταν κάτι το θετικό τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την, για την ε, Μεγάλη Βρετανία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Νορβηγίας. Ευχαριστώ. Ο Κάρολος Στάροκ για το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαι. Απαντώντας τον σοσιαλιστικό, σοσιαλιστή συναδελφό μου, καταλαβαίνω ότι η Νορβηγία έχει, ένα μεγάλο, έχει μεγάλα σύνορα, έχει μακρά σύνορα με την ε, Ρωσία και ως μέλος του ΝΑΤΟ πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την ρωσική άκτο. Εγώ σε σχέση με τον Brexit ήμουν υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δυστυχώς χάσαμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει με πιο ήπιο τρόπο αυτό το Brexit και να γίνει με, ακολουθώντας ένα μοντέλο το οποίο θα είναι Νορβηγία συν, δηλαδή να υπογράψει τη συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να διατηρήσει και άλλα θετικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά φαίνεται ότι η κυρία Μέη στην πρόσφατη της ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων λέει ότι θα είναι απότομο το Brexit, σκληρό και απότομο και κακοτράχαλο και δεν θα θέλει η Μεγάλη Βρετανία να μπει στον ε, χώρο της ΕΖΕΣ. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κατά πόσο η Νορβηγία θα χαιρόταν να ξαναγυρίσει στην ΕΖΕΣ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η Μεγάλη Βρετανία γιατί υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι μπορούσε να γίνει αυτό ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιήσει το βέτα του για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς είστε τρία μέλη και έχετε βέβαια σε διακυβερνητικό αυτό επίπεδο το δυνατότητα βέτο, αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο η Μεγάλη Βρετανία θα ανέτρεπε την ισορροπία σας. Ένα άλλο θέμα είναι η ελευθερία διακίνησης. Εσείς έχετε τονίσει ότι είναι σημαντικέ και όχι διαπραγματεύσιμε αυτέ τι τέσσερις ελευθερίες. Αλλά θέλω να ξέρω την άποψή σα, γιατί μου είπα και οι νομομαθείς ότι το άρθρο 112α της Συνθήκη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να έχει επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μονομερός να θέσει μια οροφή στον αριθμό των μεταναστών που έρχονται στην, Ηνωμένο Βασίλειο από τα 30 κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσα στα δικαιώματα που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο στην συνθήκη αυτή. Εάν και εσείς συμφωνείτε, τότε γιατί νομίζετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να ακολουθήσει την οδό του αποχωρισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Φίλε ελεύθερη. Και ο Σπέτ, ο οποίος είναι και ο εισηγητής για τα θέματα της Αρκτικής. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κύριε Μπόρκε Μπρέντε. Και είναι και πολύ κρίσιμη αυτή η στιγμή, γιατί κάνουμε και αυτή τη κοινή έκθεση για την Αρκτική. Έχω δύο ερωτήσεις να σας απευθύνω. Ε, σύντομα αναφερθήκατε στις σχέσεις σας με την Ρωσία, αλλά η αλήθεια είναι ότι πριν μερικά χρόνια, ε, η Ρωσία έχει αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές της δαπάνες για την ε, Αρκτική και ε, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τον στόχο που έχει η Ρωσία κάνοντας κάτι τέτοιο. Δεύτερον, η Κίνα, η Ινδία και κάποιες άλλες μακρινές χώρες, μακρινές από την Αρκτική, ε, δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, για την περιοχή της Αρκτική. Ε, ποια είναι η άποψη της Νορβηγίας και των γειτόνων σας επίσης σχετικά με αυτό το ε, ενδιαφέρον, το όψιμο ε, ενδιαφέρον και επίσης ποιος είναι ο αντίκτυπος που θεωρείτε ότι μπορεί να έχει σε σχέση με τους παρατηρητές τη συμμετοχή ενδεχομένως άλλων παρατηρητών στο Συμβούλιο της Αρκτικής για χώρες οι οποίες είναι πολύ μακρινές από την περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ για τους ε, πράσινους η κυρία Βαλέρο. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να μιλήσω σου και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, να μιλήσω με το γείτονά μου, τον Νορβηγό. Νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνόμαστε και καλύτερα. Ε, και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να μιλήσω ε, σουηδικά. Ναι, είναι γρήγορε πλέον οι εξελίξεις. Και ακόμα παντού, και αλλά ακόμα πιο γρήγορες ε, είναι οι εξελίξεις εις την Αρκτική. περιβαλλοντικά, ας πούμε, βλέπουμε ότι στην Αρκτική η αύξηση της της θερμοκρασίας γίνεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι σε άλλες ε, περιοχές. Επίσης έχουν ανοίξει νέες ε, ναυτικές ε, οδοί. Έχουμε επίσης το θέμα των πετρελαϊκών πόρων και της πρόσβασης κοιτασμάτων συγγνώμη, και της πρόσβασης αυτούς, αλλά δεν είναι πάντα θετικό το να ανοίγει κανείς νέες εμπορικές δραστηριότητες. Μερικές φορές είναι κακό ή εν περιπτώσει γνώση μπορεί να δημιουργήσουν ε, πολλά προβλήματα, κυρίως όταν μιλάμε για εκμετάλλευση ας πούμε αερίου ε, ή κρεσμάτων πετρελαίου που ξέρουμε ότι ευθύνονται εν τέλει για, την, ε, για το λιώσιμο των πάγων της ε, Αρκτικής. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν ε, να επιτρέψουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λοιπόν και την εξόριξη των πόρων από την Αρκτική. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την πρόσφατη απόφαση. το, ακόμα και το το, το καλύτερο πετρέλαιο κατά τη δικιά μου άποψη είναι το πετρέλαιο το οποίο έχει μείνει στη θέση του και δεν το έχει εξάγει κανείς δεν το έχει εξορίξει κανείς. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά αυτή τη χρήση των κοιτασμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω, τώρα, τώρα μπορούν να πάρουν τον λόγο εκπρόσωποι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, μάλλον ολοκληρώθηκαν ε, οι εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων, τώρα μπορεί να μιλήσει όποιο θέλει. Ε, θα ολοκληρώσω και τον κατάλογο, θα κλείσω τον κατάλογο των αγορετών έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να απαντήσετε. Τρεις ακόμα συναδέλφους. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Θα ήταν πιο εύκολο ίσως να μεταφραστούν τα πράγματα. Αν μιλούσα τη μυθική μου γλώσσα θα μιλούσα στα αγγλικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορούν να υπάρξουν εξελίξεις από τα πρόσφατα γεγονότα. Θα μπορούσε όμως η Νορβηγία να δεσμευτεί για περισσότερο ελεύθερο εμπόριο από την από στο παρελθόν με την Ευρώπη. Είσαστε βέβαια πλήρως στην ενιαία αγορά, αλλά ιδίω για τον αγροτικό τομέα θα θέλαμε η Νορβηγία να μειώσει την ε, επιβάρυνση των προϊόντων και να υπάρξει πιο έντονο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσετε να είστε με τη δική μα πλευρά στον αγώνα κατά του προστατευτισμού. επίση για τον, την περιοχή τη Ακτικής, <clears throat> Εμεί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για την Ιρλανδία. Ξέρουμε ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε και τι ε, ενέργειε έρευνα και διάσωση αν λιώσει ακόμα περισσότερο ο πάγος που καλύπτει την Ιρλανδία και αυξηθούν οι δράσεις ναυσιπλοεία στην περιοχή αυτή. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα αφήσει αυτά τα θέματα στις σκανδιναβικές χώρες ή να ασχοληθεί και η ίδια περισσότερο. την άρω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτά που είπατε. Δύο σύντομα και σημαντικά για μένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, πώς αξιολογείτε το ρόλο της Ρωσίας στην Βαλτική. Εγώ με την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συζήτηση η οποία ήταν αρκετά ανησυχητική που διοργανώθηκε από την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας με εκπροσώπους και από τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Πώς βλέπετε τη Ρωσία λοιπόν και τις εξελίξεις στη Βαλτική και δεύτερον πώς εκτιμάτε το ρόλο της Ρωσίας και τον ενδεχόμενο ρόλο τους εκεί. Και δεύτερο ερώτημα, γνωρίζοντας το ρόλο που έχει διαδραματίσει η χώρα σας ε, στην πρόσφατη ιστορία, στο να εξασφαλίσει συμφωνίες και συμφιλίωση σε πολλά θέματα Ποια θα ήταν η δική σας πρόταση για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία που γίνονται όλο και περισσότερο σχέσεις αντιπαράθεσης, σχέσεις ανησυχητικέ. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την συνέχιση της κλιμάκωσης για τις σχέσεις αυτές. Και τέλος η κυρία Φωτίγα που είναι η πρόεδρος της Υποεπιτροπής μας για ασφάλεια και άμυνα. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Είπατε τουλάχιστον δύο φορές το δίκαιο της θάλασσας σε ό,τι αφορά την Αττική. η αποστατικοποίηση συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας για την περιοχή αυτή, μάλλον η στρατικοποίηση συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας στην Αττική. Τι θα πρέπει να προβλέψουμε για τα θέματα αυτά. Και δεύτερον, έχετε κάποιες ανησυχίες για την παρουσία της ε, Ρωσίας. Βλέπετε να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις για την Ορβηγία και πόσο, σε ποιο βαθμό είσαστε διαθέσιμος να βοηθήσετε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για τη δική μου περιοχή. Εγώ προέρχομαι, όπως καταλαβαίνετε, από την Πολωνία. Ευρύ το φάσμα των ερωτημάτων. Κύριε Μπρέντε, έχετε περίπου 20 λεπτά για να απαντήσετε όλα αυτά τα ερωτήματα, τουλάχιστον όσα μπορείτε περισσότερο. Παρακαλώ, μπορείτε να παρουσιάσετε τις προτεραιότητές σας. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης ευχαριστώ και αυτές τις πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις που υποβάλλατε και μάλιστα ε, για πάρα πολλά θέματα και διαφορετικά θέματα. Επιτρέψτε μου ε, λιγάκι να τα συγκεντρώσω τα ερωτήματα. Ε, καταρχήν απευθύνομαι στην ε, βουλευτή από την Πολωνία και το θέμα της ε, ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό είναι ένα θέμα καθοριστικής σημασίας για, όλοι μας, όλους μας. Νομίζω ότι η Νορβηγία είναι ένα ιδιαίτερα προβλέψιμος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Περίπου το 25% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από την Νορβηγία. Δεν είμαι ίσως απόλυτα αντικειμενικός, αλλά πρέπει να πω ότι ο πολιτικός κίνδυνος στις εισαγωγές νορβηγικού αερίου είναι μηδενικός, ανύπαρκτος. Επίσης, με πολύ μεγάλη μας χαρά να ε, επεκτείνουμε τη συνεργασία, διότι το φυσικό αέριο είναι η γέφυρα το να περάσουμε από μια κοινωνία η οποία βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα σε μια νέα κοινωνία που θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα. Και εμείς μπορούμε να ε, αντικαταστήσουμε τον άνθρακα ε, με αέριο, γιατί οι εκπομπές διοξιδίου στο αέριο είναι οι μισέ κατά το ίμιση χαμηλότερε από ό,τι στον άνθρακα. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ε, συζητήθηκε και στην συνάντηση που έλαβε χώρα στο Παρίσι. Και αυτό έχει σχέση και με την άλλη ερώτηση που μου υποβάλλεται. Δηλαδή, αν δούμε λιγάκι το θέμα της υφαλοκρηπίδα και του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έχει όλες αυτές τις ιδιότητες που σας ανέφερα σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή διαφοροποίηση. Οι εκπομπές ε, είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι στην περίπτωση των ορυκτών καυσίμων. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ε, υφαλοκρηπίδας και να επισημάνω ότι εμείς εφαρμόζουμε τις πιο αυστηρές προδιαγρα... περιβαλλοντικές προδιαγραφές στον κόσμο. Οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα σε εμά είναι από τις χαμηλότερες στον κόσμο, ε, κυρίως ε, στην παραγωγή πετρελαίου και αερίου στη Νορβηγία. Κάτι άλλο. Το βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας, οι υδατοκαλλιέργειες και η αλληλεία, όλα αυτά μπορούν να συμβαδίζουν αρμονικά και με άλλες εξελίξεις στα ορυκτά καύσιμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, αν υπό την προπόθεση βέβαια ότι καθορίζει κανείς τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Μερικέ φορέ δεν είναι μόνο η τεχνολογία που είναι απαραίτητη, πρέπει να προχωρήσει κανείς ακόμα πιο πέρα. Εμείς, παραδείγματο χάρη, έχουμε ε, την ε, πιο καθαρή περιοχή του κόσμου από πλευράς εκπομπών και νομίζω αυτό από μόνο του είναι απόδειξη, αποτελεί απόδειξη. Με ρωτήσατε ε, για τη σχέση μας με τη Ρωσία. είναι πράγματι γεγονός το ότι υπάρχει μια ασύμετρη κατάσταση όσον αφορά στα σύνορα ανάμεσα στην Ρωσία και την Νορβηγία. Γιατί εκεί έχουμε ε, ισχυρή στρατιωτική συγκέντρωση στη Ρωσία, στο Μπυρμάνσκα και σε όλη αυτή την ε, Χερσόνησο και αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίσαμε και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Είναι λοιπόν ε, σαφές, όπως ε, υπογράμμισε και ένας ε, αξιότιμος βουλευτής, ότι πράγματι διαπιστώνουμε να υπάρχει διπλασιασμός ε, του στρατιωτικού προϋπολογισμού της Ρωσίας από το 2005 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μέσα από το ΝΑΤΟ αλλά και μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουμε το θέμα αυτό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει και να ε, βασιστούμε στην αλληλεγγύη στο ΝΑΤΟ. Αναφέρουμε συγκεκριμένα στο άρθρο 5, αριθμών 5 του ΝΑΤΟ. Πέρα από αυτό, εστιάζουμε και στο να ισχυροποιήσουμε τις ε, αμυντικές μας δυνατότητες. Όσο έχει κατάσταση ασφάλειας ε, στην ε, περιοχή που μας περιβάλλει, στην Ευρώπη γενικότερα, νομίζω το είπα αυτό στην εισαγωγική μου παρέμβαση, πλέον έχουμε μια κατάσταση όπου οφείλουμε να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες για ε, τη δική μας ασφάλεια, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ασφάλειά μας. Νομίζω αυτό έχει γίνει κατανοητό και αυτό συμβαδίζει και με τα εθνικά μας συμφέροντα. Όπως σας είπα, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά παράλληλα εφαρμόζουμε τις κυρώσεις και όλα τα άλλα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί της Ρωσίας. Νομίζω αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αντίδραση στο ότι η Ρωσία παραβίασε το διεθνές δίκαιο προσαρτώντας την Κρυμαία και επιφέροντας και αστάθεια στον Ντομπάς. Η αντίδραση ήταν κυρώσεις. Ε, αυτό λοιπόν, όπως σας είπαμε, ήταν η αντίδραση στην ε, παραβίαση των συνόρων της ε, Ουκρανίας συμφωνήσαμε με τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, νομίζω αυτό είναι γνωστό, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ε, αν κανείς θέλει να σέβεται αυτές τις δύο συμφωνίες, ε, δεν μπορεί να εισάγει κυρώσεις ε, όπως συνέβαινε μετά το ε, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η μία χώρα ε, προσαρτούσε ε, το κομμάτι μιας άλλης. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Τι είδου προηγούμενο θα προέκυπτε. Ως εκ τούτου, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτήν την κατάσταση και όπως σας είπα παράλληλα μπορέσαμε να συνεχίσουμε την προς, τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτών ε, στην Αρκτική, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον της ε, Ρωσίας. Πιστεύετε ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις και στην θάλασσα Μπάρεντς. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Εκεί μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία ε, και νομίζω ότι στο μέλλον ε, θα υπάρχει και διαφορετική στάση απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους ΛΟΑΔ ε, και ε, σε άλλα θέματα που αφορούν το Κρεμλίνο. Κατόπιν ετέθησαν ερωτήματα που έχουν σχέση με, την, με το Brexit, την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σαφήνεια για το τι θα κάνει η Βρετανική κυβέρνηση μετά την ομιλία που έκανε η κυρία η Πρωθυπουργός η Τερέζα Μέη. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία επιτιμεί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πλέον ε, θα έχει κατατεθεί και ενεργοποιηθεί το άρθρο 50. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή αυτή είναι η βάση των διαπραγματεύσεων. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει κανείς να συμφωνήσει επί της αποχώρησης και μετά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για σχέσεις ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Αν κατάλαβα καλά από την ομιλία της κυρίας Ντέβις ε, αλλά και του συναδέλφων του κυρίου Τζόνσον, του Ντέβις Ντέβις και άλλων, ε, αν κατάλαβα καλά οι Βρετανοί δεν επιθυμούν να είναι μέλος της Τελωνιακής Ένωσης ή της κοινή αγοράς. Η Μεγάλη Βρετανία επιθυμεί να έχει μια κλασική ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στην Ορβηγία, γιατί εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτής της κοινή αγοράς, άρα δηλαδή έχουμε κοινή αγορά και με τη Μεγάλη Βρετανία και πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολλές από τις δυσκολίες λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν και μας. Και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος. Ε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά συνάψει συμφωνία ελεύθερη μπορεί με την ε, Μεγάλη Βρετανία, θα το κάνουμε και εμείς. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Τώρα, ε, υποθετικές ερωτήσεις, τι θα γινόταν αν η Μεγάλη Βρετανία δεν επιθυμούσε σχέσει ελεύθερου εμπορίου. Εγώ στην πολιτική έχω μάθει ότι δεν θα πρέπει κανείς να τοποθετείται πάνω σε παραδοχές. Και επιμένω σε αυτό, ε, αν ε, αυτό είναι η επιτιμία του Ηνωμένου Βασιλείου, επ' αυτού να τοποθετηθώ. Και εγώ να σας πω ότι θα προτιμούσε σαφώς η Μεγάλη Βρετανία να έμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τη δεύτερη ή την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του, της Ευρώπης ε, προφανώς και τη χρειαζόμαστε. Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της ε, Ευρώπης. Τη χρειαζόμαστε λοιπόν τη Μεγάλη ε, Βρετανία σε αυτή την ταραγμένη περίοδο αλλά το να έχει κανείς ε, το πόδι του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, Βρετανία ε, εν περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα και θα πρέπει να σεβαστούμε το τι αποφάσισαν οι Βρετανοί Διακόπτει ο μιλητής. Eh? Ναι, ναι, μου δώσανε γραμμή να πω κάτι, λέει ο υπουργό. Για το θέμα της έκθεσης για την Ακτική. Όπως είπα και στις εναρκτηρίες μου παρατηρήσεις, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η έκθεση. Αυτή νομίζουμε ότι είναι μια εμπεριστατωμένη έκθεση και οι συμβιβαστικές ε, τροπολογίες οι οποίες έχουν τύχει διαπραγμάτευσης είναι ικανοποιητικέ. Στην Σουηδή, φίλοι μου, θέλω να πω ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι οι αλλαγές που γίνονται σε κλιματολογικό επίπεδο γίνονται με επιταχυνόμενη ταχύτητα, με διπλή ταχύτητα στην αρχική. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ. Βλέπουμε να λιώνει οι παγετώνες, το οικοσύστημα και το ενδιέτημα πολλών ε, ειδών στην Αρκτική καταστρέφεται. Λοιπόν, ανοίγει στην εκμετάλλευση η Αρκτική, αλλά ο λόγος για τον οποίο είναι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα τυχής. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και εγώ χαίρομαι που και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία συμφωνούν στο ότι πρέπει να διατηρήσουμε τους στόχους οι οποίοι έχουν <clears throat> θεσπιστεί στη συμφωνία της COP21 στο Παρίσι. Θα παραμείνουμε σε πλήρη συμμόρφωση με αυτούς τους στόχους και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων αυτών. Και μετά για το ερώτημα από τον δανόφιλο μας. για το ελεύθερο εμπόριο και για την αποτροπή του προστατευτισμού. Η κατάστασή μας αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία συνεργάζονται πολύ στενά, χάρη και μέσα από την ενιαία αγορά. Όταν ενταχθήκαμε στην ενιαία αγορά το 1992 με τη συμφωνία του ΕΟΧ, δεν γίναμε φυσικά τότε μέλη της Τελωνιακής Ένωσης. Αυτό οδήγησε και σε δυσκολίες για τις διαπραγματεύσεις ε, ένταξης της Νορβηγίας στο παρελθόν που οδήγησαν στο δημοψήφισμα του 1974. 10% του πληθυσμού μας ζει βορειότερα από τον Αρκτικό κύκλο. Ο πληθυσμός αυτός στο βόρειο τμήμα της Νορβηγίας ζει σε μεγάλο βαθμό από τη Γεωργία. έχουμε τα, τις μεγάλες πεδιάδες του βορρά με μικρά χωριά, αλλά έχουμε και ορεινή γεωργία στο, στον ακραίο βορρά της Νορβηγίας και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την παρουσία αυτών των ανθρώπων στο βορρά της Νορβηγίας. Για πολλούς λόγους είναι θετικό αυτό, για λόγους περιβάλλοντος, για λόγους ασφάλειας και όλα αυτά. αλλά δεν είναι δυνατό να μπορέσει ένα αγρόκτημα με ελάχιστα ζώα στην ε, Βόρεια Νορβηγία να συναγωνίζεται ε, τα αγροκτήματα και τις ε, εγκαταστάσεις εκτροφής στη Δανία που είναι πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανταγωνισμού. Είναι πιο οικολογικό, ίσως πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά δεν μπορεί να έχει την οικονομική βιωσιμότητα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Και αν υπάρξει κάποια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρξει μια πρόσφαση στην αγορά για τις εξαγωγές μας μεταποιημένων ηχθείων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι αποχρόντες λόγοι για τους οποίους δεν θέλουμε να συμμετέχουμε πλήρως στην Τελωνιακή Ένωση. Θέλουμε όμως παρόλα αυτά να προχωρήσουμε τι συμφωνίε του ΠΟΕ προς τα εμπρό. Γι' αυτό η Νορφηγία μαζί με την Ελβετία και ο, Κα... ο Καναδάς συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο του ΠΟΕ στην Νορβηγία, στην Αϊδόπη, συγγνώμη, πέρσι, να πάψουν να υπάρχουν πια ε, κλίμακοτα οι <clears throat> επιδοτήσεις στον τομέα της ε, γεωργίας για τις εξαγωγές. Αυτό θέτει προβλήματα για τους ε, γεωργούς μας, αλλά είναι ακριβώς το, το αποτέλεσμα των συμφωνιών του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ είναι αυτή τη στιγμή ο προμαχώνας μας εναντίον του προστατευτισμού και χρειαζόμαστε πράγματι να έχουμε πολλά τύχη και προμαχώνες σε πολλού τομεί. Θα χρειαστεί να έχουμε και τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώ, είναι έτσι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ Μπρέντε που ήρθατε εδώ στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ αξιόλογη συζήτηση λίγο πριν την ε, ψηφοφορία ε, την έκθεση για την Αρκτική που θα γίνει αύριο. Ε, θα ήθελα βεβαίως να σας συγχαρώ και σας και τη χώρα σας. Ε, κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, ε, το Σαββατοκυριακό διάβασα τον δείκτη της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εάν ξέρετε αυτό το θέμα του Democracy Index είναι, είναι μία έκθεση για την κατάσταση της δημοκρατίας σε 167 χώρες και δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Η Σουηδία είναι στην τρίτη θέση. Στη δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο, ε, είναι η Ισλανδία, αλλά για μία ακόμα φορά ε, πρωταθλήτρια είναι η Νορβηγία. Δηλαδή, για μία ακόμα φορά θεωρείται ε, η, η καλύτερη δημοκρατία υψηλότερων προτύπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Να είστε καλά λοιπόν, να τα πηγαίνετε καλά στην Ευρώπη και να συνεχίσετε αυτές τις καλές ομαλές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας. So uh, under a bit of time pressure, so we continue now and come. Πρόεδρος, συνεχίζουμε λοιπόν και θα δούμε τα θέματα 5, 6, 7 και 8 ε, που αφορούν τα Βαλκάνια. Έχουμε εκθέσεις για την Αλβανία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Μακεδονία, λέει ο Πρόεδρος, και το Μαυροβούνιο. Να δούμε λοιπόν σε δεύτερη ε, εξέταση την έκθεση για την Αλβανία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φλέγκενστάιν ε, και να μας πει δύο λόγια σχετικά με τις ε, ε, τροπολογίες και μετά θα έχουμε και κάποιες ερωτήσεις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω όμως γερμανικά. τέλη Νοεμβρίου ε, έγινε η πρώτη συζήτηση για την έκθεση και μετά κατατέθηκαν οι τροπολογίες. 231 τροπολογίες κατατέθηκαν και πρέπει να σας πω χαίρομαι πάρα πολύ που σε 18 ε, συμβαστικές προτάσεις μπορέσαμε να καλύψουμε όλες τις σημαντικές παραγράφους της ε, έκθεσης και μπορέσαμε να επιτύχουμε ουσιαστικά την πλειοψηφία και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους και ηγητές. Νομίζω με τον τρόπο αυτό ε, η έκθεση είναι και αποτελεσματική, αποκτά βάρος, δηλαδή αν ως εισηγητής μπορεί κανείς ε, να υπογραμμίσει ότι η ε, Αλβανία ε, αντιμετωπίζεται από όλε τι πολιτικέ ομάδε ε, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Η Αλβανία σημειώνει συνεχή πρόοδο στην εκπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων. Και η έκθεσή μου αναφέρει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει όταν θα έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για την δικαστική Και ε, και θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η διαδικασία εκείνη η οποία θα πρέπει να καταστήσει τη δικαστική μεταρρύθμιση αξιόπιστη. Από την τελευταία συζήτησή μας τον Νοέμβρη, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, μετά από θετική τοποθέτηση της Επιτροπής της ε, Βενετίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την συνταγματικότητα των συμφωνιών και η διαδικασία vetting στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης θα αξιολογηθούν όλοι οι δικαστές και αυτό δεν το κατάφερε μόνο η κυβέρνηση αλλά το σύνολο του Κοινοβουλίου και η αντιπολίτευση η οποία και αυτή ε, ενέκρινε αυτούς τους νόμους σχετικά με το betting, την αξιολόγηση. Ε, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, προχωράει με αργό βέβαια ρυθμό, ίσως αργότερο ρυθμό από ό,τι επιθυμούμε και υπάρχει και κάποια πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση του ε, οργανωμένου κλίματος. Ίσως όχι απόλυτα αποτελεσματική. Πρόοδος επίσης στους νόμους περί διαφθοράς και επίσης ε, και περαιτέρω εργασίες για να υπάρξει νομοθεσία σχετικά με την κατάργηση των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων. Στην έκθεση αναφέρεται το τι πρέπει να κάνει η Αλβανία. Δηλαδή να ολοκληρωθεί η δικαστική μεταρρύθμιση, να μην υπάρχουν μόνο θεαματικές ε, μεμονωμένες ε, μεταρρυθμιστικές ενέργειες, αλλά μια οργανωμένη, ένα σύστημα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου κλίματος. Και αυτό όχι μόνο κατά την ε, αστυνομική έρευνα, αλλά και κατά την καταδίκη εξόπινων πράξεων και την συντριβή των δικτύων. Αυτό που ενδιαφέρει επίση είναι να επεκτείνουμε περαιτέρω τους νόμους ε, περί διαφθοράς. Δεν έχω χρόνο. Πόσο μπορώ να μιλήσω ακόμα, λέει ο μιλητής. Μου κλέψατε 10 δευτερόλεπτα, θα επιταχύνω. Λοιπόν, θα τα λέω με λέξεις, ε, σημαντικές λέξεις. Σημαντική λοιπόν είναι η συνεργασία με κοινωνία των πολιτών, ε, τις μειονότητες, ε, ο κοινωνικός διάλογος. Υπήρξαν πολλές τροπολογίες και πολύ καλή συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ στην έκθεσή μου ε, θα ήθελα να ε, μπορούσα να μπω σε κάποιε λεπτομέρειες που δεν μπορώ να το κάνω. Θα τα πω πάλι με λέξεις κλειδί. Εξυγχρονισμός της παιδείας, ε, προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση της θέσης του διαμεσολαβητή, πολιτική ισότητα των δύο φύλων, πολιτική σταθερότητα στα Βαλκάνια. Θεωρούμε ότι η Αλβανία θα πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο που έχει ξεκινήσει. Ελπίζω να είχατε την ευκαιρία ευκαιρία να δείτε τις συμβαστικές προτάσεις. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους σκιοσυγητές. Νομίζω ότι είναι μια καλή έκθεση αυτή λόγω της αγαστής συνεργασίας που είχαμε. Ευχαριστούμε λέει και ο Πρόεδρος. Έχουμε 20 λεπτά για την Αλβανία, 1,5 λεπτό για τον κάθε σκιώδιο. Ο κύριος Κούκαν είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Φλέκενστίν για την εξισορροπημένη έκθεσή του. Εγώ υποστηρίζω τις τροπολογίες συμβιβασμού γιατί συνάδουν με την κύρια οδηγό ιδέα της έκθεσης αυτής. Πρώτα απ' όλα, δύο παρατηρήσεις. Η υποστήριξη της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας θα πρέπει να απελαμβάνει και την αναγνώριση των επιτευγμάτων της. Θα πρέπει να δώσουμε θετικά μηνύματα για να συνεχίσουν οι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη δημόσια διοίκηση και στην δικαιοσύνη και την πρόθεση των κυρίων προτεραιοτήτων. <clears throat> Επίσης μια έκκληση, μια επίγουσα έκκληση στους πολιτικούς της Αλβανίας για την προετοιμασία των γενικών εκλογών. Όλες οι συστάσεις που έχουν παρουσιαστεί για το εκλογικό σύστημα και την διεξαγωγή των εκλογών θα πρέπει να εφαρμοστούν. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί χώροι ακόμα όπου χρειάζονται Αλλαγέ ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της καλλιέργειας ναρκωτικών και της λαθεμπορίας των ίδιων αυτών. Υποστηρίζουμε επίσης την τροπολογία αυτή που είναι σημαντική για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με ορισμένα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στην Αλβανία. Είναι καλό λοιπόν να τονίσουμε και το ρόλο της Αλβανίας σε περιφερειακή συνεργασία και το τελευταίο μου σχόλιο υπάρχει και μια σειρά προβλημάτων για την προστασία των μειονοτήτων στην Αλβανία. Εγώ εντυπωσιάζομαι γιατί το θέμα αυτό δεν είχε τονιστεί τόσο πολύ από το, τους βουλευτές ακόμα και την εποχή που ήταν ο κύριος Χούντης ε, εισηγητής, ο καλός μου φίλος από την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Κούκανο, ο Charles Τένοκ. Ευχαριστώ πολύ και εμείς ως ECR ε, συγχαίρουμε τον εισηγητή για μια πολύ, την πολύ ισορροπημένη του έκθεση. Ε, η Αλβανία βεβαίως ως υποψηφία χώρα εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες ε, σε διάφορα κεφάλαια όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο συμπεριλαμβανομένο και αυτού τη δικαιοσύνη τη της του οργανωμένου εγκλήματος και κατά αυτή την έννοια θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μείζωνα προβλήματα ε, και επίσης είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την περιφέρεια και όχι μόνο των Δυτικών Βαλκανίων και όχι μονάχα την ε, Αλβανία. Ε, καλωσορίζουμε τις προτινόμενες και ε, όσον ε, ούπο ε, υποψήφιση τροπολογίες, τροποποιήσεις μάλλον του εκλογικού ε, νόμου. Είναι σαφές ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι αντιφατικά και εξακολουθούν να είναι αντιφατικά στην, στην Αλβανία, τα θέματα των αιτήσεων ασύλου κτλ. θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και θα πρέπει να δούμε και ε, μια σαφή δέσμευση όλων των χωρών αυτών στο κράτος ε, δικαίου. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά τους τζιχαντιστές από την Ιλβανία καθώς επίσης και τα μέτρα τα οποία συζητώνται και λαμβάνονται τώρα. Ίσως και ο πρόεδρος Τραμπ κάτι να καταφέρει όσον αφορά την καταπολέμηση του ISIS. Πάντως ε, είναι γεγονός ε, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν οποιοδήποτε έχουν λάβει μέρος ε, σε σκιαές πράξεις ότι θα υποστούν, θα περάσουν από δίκη. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you, Chair. Uh, first of all, ο επόμενος ομιλητής θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Φλέκενστάιν, λέει ο κύριος Κούτσουκ ε, είναι θετικό το ότι έχουν αναγνωριστεί οι πρόοδοι που έχει κάνει η Αλβανία και η αλβανική ε, κοινωνία. Ε, οι πέντε πρώτες προτεραιότητες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης αποτελούν ένα πρώτο καλό βήμα. Ε, όσον αφορά τις διαδικασίες ε, της ε, προενταξιακές. Χαίρομαι επίσης που ο κύριος Φλεκενστάιν αλλά και άλλοι συνάδελφοι συμμερίζονται την άποψή μας ότι θα είναι καλό να ξεκινήσει η ενταξιακή διαδικασία κυρίως μετά τις εκλογές. Οι δικές μας τροπολογίες αναφέρουν ότι οι επερχόμενες εκλογές του 2017 θα αποτελέσουν μια πραγματική δοκιμασία έτσι ώστε να ανοίξει η πόρτα των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ε, θα πρέπει να ε, έχουμε αυτές τις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για όλες τις άλλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Αλβανία έτσι ώστε να λάβει επιπλέον μέτρα έτσι ώστε και οι Αλβανοί πολίτες ε, οι οποίοι ε, ζουν εκτός της αλβανικής επικρατείας να έχουν τη δυνατότητα ε, να ψηφίσουν. Η τροπολογία μας γενικώ λαμβάνουν υπόψη τις, τα πολιτικά βήματα τα οποία έχει λάβει η αλμανική κυβέρνηση αλλά υπογραμμίζουν επιπλέον ότι θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα έτσι ώστε κυρίως να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευράς της ΓΚΟΕ. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φλαγκεστάιν, οι συμβαστικέ τροπολογίε που έχουν ε, προταθεί στην Επιτροπή καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα μεγάλα ζητήματα τη έκθεση. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να σταθώ σε δύο θεμελιώδη ανταξιακά κριτήρια που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, αλλά ιδιαίτερα κατά την ενταξιακή διαδικασία, θα γίνονται απόλυτα σεβαστά από τις χώρες. Το πρώτο έχει να κάνει με τον πλήρη σεβασμό των μειονοτήτων και το δεύτερο με την ανάπτυξη και την διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται και στη φετινή έκθεση, η Αλβανία θα πρέπει να εργαστεί όπως οφείλει για τη βελτίωση των συνθηκών όλων των μειονοτήτων στη χώρα και ενώ αναφέρεστε σε άλλε μειονότητε, παραδείγματο χάρη του Ρωμά, δεν αναφέρεται τίποτα για την ελληνική μειονότητα, όπως δεν αναφέρεται και τίποτα για την υποχρέωση της χώρας να ενισχύσει όπως οφείλει το νομικό καθεστώς που διασφαλίζει την προστασία των μειονοτήτων και ιδιαίτερα την προστασία του δικαιώματος στην διοκτησία. Δεν θέλω να αναφέρω το περιστατικό, το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Θέλω όμως να τονίσω εδώ ότι ο συνήγορος του πολίτη στην Αλβανία, το σχετικό πόρισμα που, στο σχετικό πόρισμα που εξέδωσε, ζητά από τις αλβανικές αρχές τον αυστηρό σεβασμό της νομικής διαδικασίας, η οποία έχει παραβιαστεί ως προς την έγκριση σε του σχεδίου ανάπλαση τη χυμάρα και την αναστολή κάθε παραπέρα ενέργεια στην εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου ανάπλαση. Κλείνοντα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ενώ προσθέθηκαν αναφορέ για την διασφάλιση και της προόδου στη σχέση καλή γειτονία, η τελευταία πρόταση τη συμβαστική τροπολογία 18 κακώ εξισώνει τι ευθύνε των δύο πλευρών ε, και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρο ότι είστε ενήμερο ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έξαρση αλυτρωτικών αναφορών από την, πλευρά, τόσο του Αλβανού Πρωθυπουργού όσο και από τα μέλη τη κυβέρνησή του εναντίον τη χώρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νέσεριτς για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και θέλουμε να Θέλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Φλέκενστάιν για την πολύ καλή του έκθεση. Ο τρόπο που διαχειρίστηκε όλο αυτό το θέμα ήταν θετικό, ήδη το σχέδιο έκθεση ήταν πολύ θετικό και οι συμβαστικέ λύσει που επιτύχαμε είναι πάρα πολύ καλέ, πιστεύω. Και υπήρξε μια υποστήριξη σε όλε από αυτέ από του πράσινου. Δύο σημεία μονάχα για το περιεχόμενο. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας <clears throat> στην τροπολογία 168 η οποία ε, αναφέρει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βεντέτες στην Αλβανία, κάτι το οποίο αναφέρει και η έκθεση της Κομισιόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε πολλά προβλήματα για πολλές οικογένειες και παιδιά, ακόμα που κινδυνεύει το δικαίωμά τους για τη ζωή και την παιδεία στην Αλβανία. Και επίση θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Κούκαν για τη θετική γλώσσα που έχουν για την υποστήριξη των υδροηλεκτρικών έργων και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε μια καλή συμβαστική λύση στην τροπολογία 16, αλλά να υπογραμμίσω ότι από τα 71 υδροηλεκτρικά αυτά φράγματα, 44 είναι σε προστατευμένε περιοχέ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει η αλβανική κυβέρνηση. Εμεί χαιρετίζουμε λοιπόν τη στάση της Αλβανίας για τη δημιουργία εθνικών δρυμών, αλλά θα θέλαμε να ε, καλύψει όλο το, όλες τις ποτάμιες περιοχές στην Αλβανία. Ευχαριστώ. Τέσσερις ακόμα ομιλητές. Αν παραμείνετε σε ένα λεπτό ο καθένας, είναι εφικτό να το κάνουμε αυτό. Η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλέκενστάιν για αυτή την έκθεση και ιδίω για τι τόσο επιτυχεί τροπολογίες συμβιβασμού. Μπορούμε να βρούμε ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδο στου πέντε κέριους τομεί. Εγώ θα ήθελα να σταθώ προς στιγμή στο θέμα του περιβάλλοντο. Έχουμε προβλήματα όχι μόνο εσωτερικού χαρακτήρα με τους υδάτινους πόρους στην Αλβανία, αλλά υπάρχουν και προβλήματα στην Αδριατική που έχουν και επίπτωση στην Κροατία. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι οι καλές γειτονικέ σχέσεις και η περιφερειακή συνεργασία είναι θετικές, αλλά στην αρχή αυτού του μήνα υπήρξε μια ε, κοινή ενέργεια με την Κροατία και το Μαυροβούνιο και την Αλβανία που ήταν θετική και υπάρχουν επίσης και προτάσεις για τη δημιουργία αγωγών φυσικού αερίου στην περιοχή. Ο κ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Αυτοί, αυτές οι χώρες τις οποίες ε, ε οι οποίες, στις οποίες αναφέρονται εκθέσεις μας δείχνουν ότι πολλές φορές ε, είμαστε άδικοι ε, με κάποιες χώρες. Ε, ερωτώ, η Αλβανία έκανε προόδους, ναι και πολλές. η Αλβανία παίζει επικοδομητικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο, βεβαίως και αυτός ο ρόλος αναγνωρίζεται η, ε, η στήριξη όλου του πολιτικού τόξου ε, των, ε, στις πολιτικές ε, και πολιτικές μεταρρυθμίσεις ε, υπάρχει στα τύρανα, ναι, υπάρχει και επομένως αν θέλουμε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει, θα πρέπει να ανοίξουν κάποια κεφάλαια. Ξέρω ότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τώρα την Αλβανία έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρους από το ECR. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Θα έπρεπε να έχω περισσότερο από ένα λεπτό στη διάθεσή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με ξεχάσατε πριν. Αυτά που περιγράφονται Συνεχίζω ελληνικά. είναι πάρα πολύ καλά και η έκθεση είναι σωστά δομημένη, αλλά πιο πολύ εκφράζουν ευσεβείς, ευσεβείς πόθους παρά την πραγματικότητα είναι γεγονός ότι η διαφθορά, η κακή διοίκηση, δεν υπάρχει καθόλου χρηστή διοίκηση σε αυτή τη χώρα. Ε, η εγκληματικότητα είναι παντού και πολλοί εγκληματίες έχουν κέρυες θέσεις στην δημόσια διοίκηση. Το να λέμε ότι έχει κάνει πρόοδους, ναι, έχει κάνει πρόοδους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που να τις δίνουμε και εύσημα για την προκοπή που έχει κάνει. Όσον αφορά τις μειονότητες, Πέρασα αρκετές μέρες με την ελληνική μειονότητα στις μειονοτικές περιοχές και πραγματικά αυτά που έχω ζήσει δεν μπορούν να περιγραφούν ούτε σε ένα λεπτό ούτε σε μία ώρα. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ε, Ελλήνων της ε, Αλβανίας, οι μετακινήσεις πληθυσμών στις νότιες περιοχές, μουσουλμανικών πληθυσμών, οι διαφοροποιήσεις των διοικητικών ορίων των Δήμων προκειμένου να μην εκλέγεται Έλληνας εκεί που θα μπορούσε να εκλεγεί, η καταπίεση της εκπαίδευσης και του θρησκευτικού αισθήματο και κυρίως η, κατα... η παραβίαση του δικαίωματος στην ιδιοκτησία είναι σημεία τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε κατά τη δικιά μου εκτίμηση μια ad hoc επιτροπή να τα, να τα δει και να επισκεφτεί αυτή την περιοχή της χώρας. Σας ευχαριστώ. Thank you. And finally, for one minute, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Φικενστάιν για την ισορροπημένη έκθεση που παρουσίασε. Μας ανέφερε τις πρόοδους που έχει σημειώσει η Αλβανία, επίσης ανέφερε και τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να προσεχθούν και να υπάρξει σε αυτά πρόοδος, τόσο ώστε ε, να γίνει εφικτή η έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων των ενταξιακών. Ε, δεν αναφέρθηκε βεβαίως όπως ε, προείπαν και οι δύο προλαλήσατε συνάδελφοί μου, δύο προλαλήσασες συνάδελφοί μου, για, τα, για την καταπίεση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί είναι το γεγονός ότι η Αλβανία είναι η μόνη από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εκφράζει επικρατικές βλέψεις και αλυτρωτισμό για όλες τις γειτονικές της χώρες. Με κυρία προσπάθεια προς την Ελλάδα έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη στο τι ε, παραβιάσεις των συνθήκων καλής γειτονίας κάνει η Αλβανία. Πρέπει λοιπόν να μην αρχίσουμε τι ε, διαδικασίε Εντάξει, αν προηγουμένω δεν σημειωθεί πρόοδο και σε αυτά τα σημεία, γιατί τότε θα έχουμε ε, μια ανάλογη κατάσταση με αυτή που βλέπουμε με την Τουρκία. Δηλαδή, να συνομιλούμε παρά το γεγονό ότι δεν υπάρχει πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλέκενστάιν, θέλετε να, δώσετε κάποιες απαντήσεις, σε συντομία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία σημεία και μόνο θέλω να αναφέρω για να εξοικονομήσω και λίγο χρόνο. Ναι, πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι σύμφωνοι οι Έλληνες συνάδελφοι για κάποια σημεία, γιατί δεν προσπάθησα να μπω σε ειδικά προβλήματα με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά έκανα μια γενικότερη ε, διατύπωση. Υπάρχουν και άλλες βέβαια μειονότητε όμως για τις οποίες είναι απαραίτητη η βελτίωση τη κατάστασή τους. Δεύτερον, η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ποιο βαθμό μπορούμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά θέματα της Αλβανίας. Εμεί μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της ε, Αλβανίας και από την άλλη μεριά βέβαια είναι κρίμα όταν ε, ακολουθείται μια πολιτική η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για το περιβάλλον. Και τέλος το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι επαγγελματικές δυνατότητες για τους νέους στην Αλβανία. Εκεί πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στο μέλλον γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα και αυτό αυξάνει και τι αιτήσει ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται περισσότερα πράγματα στι χώρε αυτέ και στην Αλβανία συγκεκριμένα για να βοηθήσουν του νέου ανθρώπου. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρο, δεν υπήρξαν ειδικά ερωτήματα προ τον εκπρόσωπο τη DGNIR. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, εκτό αν έχετε αντίρρηση. Ωραία, τότε αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 31 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ για την συμβολή όλων σας και προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι <clears throat> το σημείο 6 η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 που αφορά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είμαστε στη δεύτερη εξέταση αυτής της έκθεσης και με χαρά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντάν Κρίσιαν Πρέντα. Τρία και μισό λεπτό έχετε κύριε Πρέντα, όπως και ο κύριος Φλέκερστάιν προηγουμένως. Τρία λεπτά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που, ε, με τους οποίους συνεργάστηκα φέτος. 288 τροπολογίες ε, είχαμε. Μέσω των ε, τροπολογίων μέσω των 153 συμβαστικών τροπολογιών προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Το κύριο μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε είναι ότι υποστηρίζουμε την Βοσνία Ριζεγοβίνη στην, ε, στην ε, ενωσιακή ε, ενταξιακή της πορεία και ότι θέλουμε να τους στηρίξουμε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει και οπωσδήποτε οπωσδήποτε θα πρέπει να προωθηθούν ε, όλες αυτές ε, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί. Ε, επίσης αναφερόμαστε στα θεσμικά, στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και εκφράζουμε τη λύπη μας διότι υπάρχουν πολιτικά και άλλα ζητήματα τα οποία με κακό τρόπο επηρεάζουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Επίσης, καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίση, υπογραμμίζουμε κάτι το οποίο είναι γνωστό σε όλου, ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αποτελεσματική χώρα, ε, θα πρέπει να βασίζεται στο, ε, στο, στο κράτο δικαίου και στο, στην ισότιμη ε, εκπροσώπηση όλων. Επίση, θα, θα πρέπει να καταγραφούν αρχέ οι οποίε από τι οποίε μάλλον θα απορρεύσουν οι μεταρρυθμίσει. Ε, όσον αφορά την νομιμοποιημένη εκπροσώπηση κτλ. Αυτό ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ε, δημιούργησε έτσι μεγάλη ανησυχία σε κάποια πολιτικά κόμματα της Βοσνίας. Ήμουν ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα εκεί ε, και ε, προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τους διάφορους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για να συζητήσω μαζί τους. Επίσης πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Σαράγεβο συζητήσαμε και με τους συναδέλφους από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας Δίας Ερζεγοβίνης. Έχουμε εδώ ε, μια συμβαστική η οποία αφορά ένα πολύ θερμό ε, θέμα, δηλαδή ε, όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης που έπρεπε να είχαν ήδη πριν από 18 μήνες εγκριθεί. Είναι πραγματικά και θέλω να το πω και να το τονίσω εδώ, είναι κρίμα, είναι ντροπή που στην ε, στο Κοινοβούλιο της ε, Βοσνίας ε, δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή για την καλή λειτουργία και τους κανόνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τη Βαζία Ριζαγοβίνη. εάν η ίδια η Βουλή δεν ενδιαφέρεται να μας ε, συναντήσει και χρησιμοποιεί κάθε μέσο έτσι ώστε να μπλοκάρει την συνάντησή μας. Επίσης, ήθελα να πω ότι έχουμε το συμβιβασμό 20 ε, που αφορά την ελευθεροτυπία, την ελεύθερη ε, έκφραση γνώμης από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι και αυτό ένα ενσυχητικό θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα εμείς είπαμε ότι θα πρέπει ανεξάρτητα ο τύπος να κάνει τη δουλειά του και χωρίς καμία παρέμβαση από πλευρά του πολιτικού κόσμου. Αυτά ήθελα να σα πω και σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Merci. Thank you. That was exactly three and a half minutes. Excellent. And now I give the floor to Mr. Pizzula, who of course is the chair of our parliamentary delegation with Bosnia and Herzegovina. Hvala. Želim prije svega čestitati kolegi Predi na odličnoj suradnji na ovoj rezoluciji. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Πρέντα για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε για αυτή την έκθεση γιατί είναι πολύ πολύπλοκη η πολιτική κατάσταση στη Βοσνία ζεγοβη Είναι δύσκολο να φανταστούμε κάτι πιο πολύπλοκο και είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας με αυτή τη χώρα. Η έκθεση αυτή λοιπόν είναι μια ευκαιρία <clears throat> να θέσουμε το ερώτημα στους εαυτούς μας ποια είναι η πραγματικότητα στη Βοσνία ζεγοβη Έχουμε υπόψη μας βέβαια τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν στη Βοσνία Ζεγοβίνη για θέματα ασφαλείας, αλλά κυρίως το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή είναι εσωτερικής πολιτικής φύσης. Υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις της Βοσνίας Ζεγοβίνης που έχει συνάψει για να προχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω πρόθεσμα και πρόθεσμα αλλά απαραίτητο είναι να υπάρξει και μια μεταρρύθμιση της συμφωνίας του Ντέιτον. Οποιαδήποτε λοιπόν μελλοντική λύση μπορεί να βασιστεί σε εσωτερική συνένεση και βέβαια δεν μπορεί να επιβληθεί εκ των έξω. Κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι όλα τα συνιστόντα έθνη θα πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους και αυτό θα πρέπει να περιλάβει και όλες τις μειοψηφίες, τις μειονότητες μάλλον. Και όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη Βοσνία-Ζεχοβίνη δεν πρέπει να το πράξουν. Και το βασικό ερώτημα είναι ποια θα είναι και η θέση τη νέα Αμερικανική διοίκηση εναντί των Βαλκανίων. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Ερχόμαστε στου ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Πρώτος, η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Σουίτσα. Συγγνώμη. Ο κύριος Παπαδάκης πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε υπόψη του αρκετέ από τι τροπολογίε μου στου συμβιβασμού και κυρίω για την έφαση στην κοινωνική διάσταση που παρότι αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανανεωμένης προσέγγισης της Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έλαβε μέχρι σήμερα την αναγκαία προσοχή. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να μην στείλουμε λαθασμένα ή μη ξεκάθαρα μηνύματα που θα μπορούσαν άθελα μας να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση σε μια πολύπλοκη και διχασμένη χώρα. Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι στην αναφορά και προώθηση της έννοιας των ίσων δικαιωμάτων για τους συστατικούς λαούς Constituent Peoples στην τροπολογία 2. Το ερώτημα που θέλω να θέσω σε όλους αυτήν την αίθουσα, το οποίο θα θέσω και αργότερα στα πλαίσια συζήτησης της δικής μου πολιτικής ομάδας, πρέπει να είναι ποιος είναι ο στόχος μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουμε την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ζητούν ίσα πολιτικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες της χώρας ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση και έτσι να στηρίξουμε την προσπάθεια σταδιακής δημιουργίας μιας κοινή πολιτιακής συνείδησης ή να ξανατονίσουμε και ενδεχομένω να υποστηρίξουμε τον περαιτέρω πολιτικό και πολιτιακό διαχωρισμό. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον πρώτο δρόμο. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να επανεξετάσει τον συμβιβασμό και να τον αναδιατυπώσει στη βάση της δικής του αρχικής τροπολογίας 77 και της πανομοιότυπης δικής μου τροπολογίας 232, οι οποίες ζητούν το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της χώρας, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε κάποιο συστατικό λαό ή όχι. Φυσικά θα τον κρατήσω ενήμερο για τη σχετική απόφαση της πολιτικής μου ομάδας αργότερα απόψε. Ευχαριστώ. Thank you. Next. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ράντος, εκ μέρους της ε, Άλντε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα και τους υπόλοιπους σκιώδησηγητές ε, γιατί πραγματικά έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Η έκθεση παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βοσνία Ερσεγοβίνη. Οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Η Βοσνία Ερσεγοβίνη αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων και το θέμα είναι πώς ε, θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και επίσης ε, και πώς θα λειτουργήσουν οι μηχανισμοί συντονισμού. Αυτό παίζει ρόλο, είναι πώς θα λειτουργήσει το μέλλον αυτή η χώρα με τις πολλές ασυμμετρίες. Ε, πράγματι πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Η Βοσνία Ερσεγοβίνη βασίζεται σε μια διεθνή συμφωνία σε σχέση με το Σύνταγμα της. Η Αμερική και η Ρωσία είναι οι χώρες που οδήγησαν στη Συμφωνία της Βοσνίας Ευθυγωπίνης και είναι δύσκολο να λειτουργήσει αυτή η Συμφωνία. Το, η δική μας έκθεση δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δύσκολα τα πράγματα στη Βοσνία Ευθυγωπίνη. Το ένα κομμάτι της <coughs> χώρας αμφισβητεί συνεχώς την βιωσιμότητα του κράτους. Ε, μιλάμε όμως για Ευρώπη. Ως εκ τούτου ε, η ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να ασχοληθούν περισσότερο με την Βοσνία Ερσεγοβίνη, όπως βεβαίως και περισσότερο και με τα Βαλκάνια γενικότερα. Ο κύριος Μέζαρετς από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, αλλάζω ιδιότητα. Ο συνάδελφός μου που θα μίλαγε κανονικά ε, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα στη Σλοβενία Ω ε, ως εκ τούτου μεταφέρω το δικό του το μήνυμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πρέντα και άλλους συνεισηγητές για τη σκληρή δουλειά και τη συνεργασία. Η Βοσνία Ερσεγοβίνη είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, ε, έλλειψη ελευθερία τύπου, υψηλή ανεργία, οικονομικά προβλήματα. Αυτά οδηγούν ε, σε αφέμαξη εγκεφάλων, πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του ψηφίσματος. Ε, με τους και οδησηγητές μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Ε, χαιρετίζω την προσέγγιση του κυρίου Πρέντα, θέλει να παραμείνει θετικός ε, σε όλο το ψήφισμα παρά τις σχολείς που αντιμετωπίζει η Βοσνία Ερσεγοβίνη. Δυστυχώς όμως κάποια εθνικιστικά συμφέροντα επικράτησαν και μπόρεσαν να επιβάλλουν κάποιες λέξεις που εμείς όμως δεν στηρίζουμε. Αναφέρομαι στη συμβαστική 2-2 του αρχικού κειμένου. Είναι μια συμβαστική πρόταση η οποία τονίζει τη διάσταση την εθνοτική στη χώρα και ε, εμείς είμαστε υπέρ της ομοσπονδιακής ε, διακυβέρνησης. Αυτή η τροπολογία είναι απαράδεκτη για μας. Ε, σας είπα ότι δεν χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει στην παλαιότερη προσέγγιση του, γιατί ε, δεν βοηθάει. Εμείς ε, ως πράσινοι πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμε ανάμεσα στους λαούς ε, της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εξάλλου αποφανθεί επίσης επ' αυτού και ολοκληρώνοντας Θέλω να πω ότι αν τελικά ε, κατατεθεί αυτή η τροπολογία, δεν θα τη στηρίξουμε. Thank you. We have three more colleagues who would like to say something. If everyone keeps to one minute. Λοιπόν, να πω, λέει ο Πρόεδρος, ότι ε, αν έχει την καλοσύνη να, να τηρείτε το χρόνο, το ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω πράγματι να παραμείνω στο ένα λεπτό. Θα ήθελα ε, να κάνω ακριβώς το αντίθετο ε, και να συγχαρώ τον κύριο Πρέντα γιατί χρησιμοποιεί μια πολύ σαφή γλώσσα και δεν αμφισβητεί τα επιτεύγματα όπως ε, είναι επικουρικότητα. Ε, όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας ε, και όσον αφορά τις προκλήσεις της εσωτερικής πολιτικής, νομίζω ότι μεγάλη επιρροή ε, ασκείται στη χώρα και οι τρεις συνιστώντες λαοί νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσοι, κυρίως οι Κροάτες, ε, διότι οι ε, Κροάτες ε, δυστυχώς δεν μπορούν να σκίσουν τα δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί από πολλές συμφωνίες, κυρίως από τη συμφωνία του Ντέιτον. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να παραμελούμε τα Δυτικά Βαλκάνια, πρέπει να παραμείνουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Ο κύριος Τάνοκ παρακαλώ για να λεπτό. Και εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πρέντε γιατί πράγματι πάντα είναι μεγάλη η πρόκληση να αναφέρεται κανείς κάθε χρόνο για την Βοσνία Ερσεγοβίνη. Από τον Τέιτον έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία και εξακολουθεί να υπάρχει μία κατάσταση όπου η χώρα δεν λειτουργεί ε, τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε. Ε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχουν αποσπαστικές ε, δυνάμεις. Έχει βάλει το δάκτυλό της και η Ρωσία. Υπάρχει μία περίπτωση επί της οποίας αποφάνθηκε το δικαστήριο και η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία. Εν πάση περιπτώσει, η Βοστιά Ερσεγοβίνη έχει καταθέσει μια αίτηση για να εξεταστεί από το Συμβούλιο. Και ελπίζουμε ότι θα εξεταστεί σωστά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι του χρόνου τέτοια εποχή ίσως η Βοστιά Ερσεγοβίνη να είναι υποψήφια χώρα. Αλλά Μέχρι τώρα, εκτός από τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και το Κοσοπέδιο, όλες οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι υποψήφιες χώρες. Ίσως και αυτή μπορεί κάτι να κάνει για να προχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ζελίμοβιτς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την εντυπωσιακή του δουλειά. Είναι δύσκολο να τοποθετείται κανείς επί του θέματος. Βέβαια το Κοινοβούλιο αποτελείται από αρκετές ομάδες και τελικά όμως φοβάμαι ότι στέλνουμε αντιφατικά μηνύματα. Να επισημάνω δύο. Το ένα είναι ότι μιλάμε κατ' ουσίαν για την αναγκαιότητα η χώρα να έρχεται στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο με μία φωνή. Από την άλλη, το λέμε αυτό, από την άλλη όμως επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ομοσπονδιακή μορφή που στη Βοσνία σημαίνει εθνοτική ομοσπονδιοποίηση κάτι που θα δημιουργούσε μεγαλύτερη διαίρεση και διχασμό στη χώρα και μεγαλύτερη δυσλειτουργία λέμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το Σύνταγμα, η Συμφωνία του Ντέιτον που ξέρουμε πολύ καλά είναι εκείνη που κρατάει τη χώρα ενωμένη. Από την άλλη όμως υποβάλλουμε αιτήματα που κατ' ουσίαν αμφισβητούν τη Συμφωνία του Ντέιτον. Και θέλω να συνεχίσω στη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρέντα. Να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή πορεία αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και έχουμε τον ε, ε, την ε, κυρία Σόφκο, η οποία ε, έρχεται η ίδια από τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να πω ότι ε, είμαι κροατίσα από την Βοσνία της Έχω ζήσει τα προβλήματα όλα αυτά ε, από πρώτο χέρι. Καλωσορίζω την έκθεση του κυρίου Πρέντα, η οποία πραγματικά θέτει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων των προβλημάτων της ε, Βοσνίας της το 2014 και το 2015 το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ε, τις βασικές αρχές της ομοσπονδιοποίησης που είναι ο μόνος τρόπος ε, σεβασμού ε, της συστατικής αρχιτεκτονικής της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, βεβαίως πολλά καλά ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι που όμως ε, ίσως αναφέρονται σε έναν ιδεατό κόσμο. Μετά από τον πόλεμο στη Βοσνία Ζεγοβίνη μάθαμε ότι πρέπει να μάθουμε τα διδάγματα του παρελθόντος ε, και να προσπαθούμε να βρούμε πρακτικές βιώσιμες ε, λύσεις και όχι να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες ε, είναι αδύνατον ε, να υλοποιηθούν. Έχουμε ε, Βοσνίους, Κροάτες και Σέρβους στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Θα πρέπει οποιαδήποτε λύση να σέβεται και τις τρεις εθνότητες και ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα προχωρήσει σωστά η συζήτηση και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συνάδελφε Ζόφκο. Κύριε Πρέντα, θέλετε να πείτε δύο λόγια ολοκληρώνοντας. Η Κομισιόν, α, η Κομισιόν δεν αναφέρθηκε ρητά, αλλά από ό,τι φαίνεται θέλει να πει κάτι. Ε, ωραία, ναι, ναι, θέλω να πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα λοιπόν και εγώ θα είμαι πάρα πολύ ε, σχετικά με τον όρο constituent people και την... And ε, as it has been pointed out, it has led to συνιστώντες λέει στα ελληνικά και σχετικά ε, με, την, ε, ε, το εθνοτικό υπόβαθρο το οποίο υπάρχει και με βάση τις αποφάσεις του Σίντιξη και του Φίντσι είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτιακή συνοχή της ε, ε, χώρας ε, γιατί οι αρχές του Dayton ήταν καλές έτσι ώστε να σταματήσει ο πόλεμος αλλά θα πρέπει τώρα να προχωρήσουν τα πράγματα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με το ενωσιακό κεκτημένο. Ευχαριστώ πολύ και τέλος κύριε Ισηγητά θέλετε να ολοκληρώσετε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς που έλαβαν το λόγο. Να σας πω καταρχήν ότι λυπάμαι για το γεγονός ότι όταν επισκεφθήκαμε το Σεράγεβο δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε την κυρία Τζένοβιτς η οποία θα πρέπει και αυτή να συμπεριλάβει και τη Ρεπούμπλικα Σύρφσκα στη διαδικασία αυτή. Και ένα δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω αναφέρθηκε το θέμα της, ε, των Πολιτειών, Μα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις Πολιτείες. Πρέπει να παραμείνει λοιπόν σε συμφωνία με αυτό το οποίο κάνουμε και εμείς. Η αμερικανική παρουσία θα ήταν ανόητο να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους Αμερικανούς στη Βοσνία. Τρίτο σημείο. Ελπίζω πράγματι ότι οι συνάδελφοί μας από τη σοσιαλιστική ομάδα θα υπερψηφίσουν τις συμβαστικές τροπολογίες Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν μια, να υπάρχει μια πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Συντηρητικών και των Φιλελευθέρων, που είναι αυτή που εξέλεξε και το νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εγώ προσβλέπω και στη συνεργασία με τους σοσιαλιστές και αυτό που ελαμβάνει και τους συνιστώντες λαούς, κάτι το οποίο έχει αναφερθεί σε όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά μας. Πρέπει να σας πω ότι από αυτή τη συνεδρίαση ήμουν παρόν σε μια συνεδρίαση της ε, συνταγματική Επιτροπής. Ένα από τα προβλήματα που συζητήθηκε εκεί ήταν η κατανομή των αρμοδιοτήτων μετά το Brexit. Η Βοσνία Ζεγοβίνη αναφέρθηκε ως μια χώρα η οποία μπορεί να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 11 κοινοβούλια. Εδώ λοιπόν ζητώ από τους σοσιαλιστές να σταματήσουν τον πόλεμο που άνοιξαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Βοσνίας και, της, και το αντίστοιχο της Κροατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέγει ο πρόεδρος. Η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί επίσης αύριο, όπως ξέρετε. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 7, την έκθεση για την ε, πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρώτη φορά που εξετάζουμε αυτήν την έκθεση που αφορά την μου ε, για το 2016 και όπως είναι η καλή παράδοση στην Επιτροπή μας θέλω να ξεκινήσω με τον εισηγητή, τον κύριο Ιβο Βάιγκλ για μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεώς του. Πόση ώρα? Έχουμε μισή ώρα για το θέμα αυτό. Θα έλεγα Πέντε λεπτά σας φτάνει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όχι, όχι. Είναι η πρώτη εξέταση της έκθεσης. Πέντε λεπτά λοιπόν για αυτό το λόγο. Είμαστε πολύ γενναιόδοροι όταν βρισκόμαστε εδώ στα πάνω έδρανα. Ευχαριστώ λέει κύριος Βάγγελ. Δεν θα σας κάνω τώρα μία σύνοψη της έκθεσης, την έχετε πάρει όλοι σας, την έχετε στους φακέλους σας. Θα ήθελα να ακούσω όμως τα δικά σας σχόλια περισσότερο. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να ακούσω τα δικά σας σχόλια, γιατί τα δικά μου σχόλια τα έχετε διαβάσει. Απλώς θέλω να πω το εξή. Το κέριο θέμα, όταν μιλάμε για την πρώην Οικοσλοβική Δημοκρατία τη Μακεδονία είναι <clears throat> το αν θα επιτρέψουμε στη χώρα αυτή να μπορέσει να προοδεύσει προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή αν η χώρα αυτή θα παραμείνει στάσιμη εκεί που βρίσκεται σήμερα, στον προθάλαμο, στον θάλαμο αναμονής για τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η χώρα αυτή εδώ και πολλά χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή η χώρα εκπληρεί τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου περισσότερο από όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες, αλλά αυτό δεν ήρκεσε για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Εφέτος, η Κομισιόν έθεσε σε εξάρτηση την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την επίτευξη των, με τη διενέργεια μάλλον των ε, πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών. Για πρώτη φορά έγινε κάτι τέτοιο. Οι εκλογές όμως αυτές έγιναν διενεργήθηκαν με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, με ίσονες ατασταλίες, χωρίς μεγάλα προβλήματα, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή η δημοκρατία, η δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει ακόμα κυβέρνηση και η διαδικασία δημιουργίας κυβέρνησης είναι αρκετά πεπλεγμένη. <clears throat> Στα Σκόπια εξετάζονται διάφορες εναλλακτικέ λύσεις και η λιγότερο ελκυστική λύση και η λιγότερο αποδεκτή για τη μελλοντική σταθερότητα της χώρας αυτής είναι η επιλογή του να επαναληφθούν οι εκλογές. Αλλά αν επαναληφθούν οι εκλογές, αυτό θα σήμαινε ότι η κρίση η οποία σοβεί στην χώρα αυτή θα συνεχιστεί και αυτό σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να μπορέσουμε να, να, να υπάρξει η συμφωνία του Μπόρζιν, όλα αυτά θα είναι επιματέο. Και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη συμφωνία είναι σημαντικές. Λένε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να φροντίσουν ώστε κατά προτεραιότητα να θέσουμε τα κρατικά συμφέροντα και όχι τα δικά τους τα στενά κομματικά συμφέροντα. Μια δεύτερη σημαντική πτυχή της συμφωνίας του Πόρζιν είναι η δημιουργία ενός Υπουργείου, μάλλον ενός ειδικού εισαγγελικού γραφείου που θα ασχοληθεί με το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Και επίσης θέλουμε να τονίσουμε και ορισμένα περαιτέρω σημεία. Το ρόλο της χώρας αυτής μέσα στη μεταναστευτική κρίση στα... οι προσπάθειες της χώρας αυτής για τη σταθεροποίηση της σύνολης περιοχής, η συνεργασία της με διεθνείς αποστολές και ενέργειες. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και πολλά αρνητικά στοιχεία, όπως η συνεχιζόμενη διαφθορά. Η έλλειψη σεβασμού των ικανοποιητικών ε, καθοποιητική προστασία των μειονοτήτων και η μη εφαρμογή σε πλήρε επίπεδο συμφωνία τη Αχρίδας 2. Όλα αυτά γεννούν μεγάλα ερωτηματικά. Επομένω, η πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία χρειάζεται την υποστήριξή μα, δεδομένου κιόλα ότι αγωνίζεται για τη σταθερότητα όλη αυτή τη περιοχή. Η χώρα αυτή, λοιπόν, <clears throat> θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει έναρξη των διαπραγματεύσεων, γιατί αυτό είναι πρωταρχική σημασία για τη χώρα αυτή. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να υπόκειται η έναρξη των διαπραγματεύσεων στην επίλυση διμερών θεμάτων, όπως είναι το θέμα του ονόματος της χώρας αυτής. Και η Κομισιόν θα πρέπει με πιο ενεργό τρόπο να προχωρήσει για την επίλυση του ζητήματος που έχει να κάνει με το όνομα της χώρας αυτής μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς και τα Ηνωμένα Έθνη. Το θέμα αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιληθεί οριστικά. Ευχαριστώ πολύ. Και σας γλίτωσα και ένα λεπτό που θα δώσω στον κύριο Φλέκενστάιν. Thank ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο ε, της ε, εκπροσώπης της ε, ΦΥΡΟΜ, τον κύριο Πίτελα, Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε αυτά που ο εισηγητής κύριος Βάιγκελ ανέφερε. Νομίζω ότι η προσέγγιση είναι αισιόδοξη και επομένως ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας που αναφέρατε ε, μπορώ να πω ότι αυτή η χώρα ε, ως υποψηφία χώρα έχει ε, κάνει πρόοδους έχει καλύψει κάποια από τα στοιχεία της συμφωνίας του Προζίνο, ωστόσο παραμένουν κάποια σημεία προς επίλυση. Επίσης, Επίσης ε, θα πρέπει να βρεθεί και κάποιος ε, πολιτικός εκπρόσωπος ο οποίος ε, θα είναι αυτός ο οποίος θα θεθεί επικεφαλής της κυβέρνησης του της, της χώρας διότι θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα και προς συμφέρον βεβαίως της ίδιας της χώρας να υπάρξει κυβέρνηση. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι περίπλοκη. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία οδήγησε σε μεγάλο μπλοκάρισμα ε, στην χώρα αυτή και επομένως το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι εν τέλει μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ε, που εξακολουθεί η χώρα να έχει ε, την δυνατότητα ε, να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις όταν και εφόσον οι προϋποθέσεις ε, καλυφθούν. Επομένως θα πρέπει η ίδια η χώρα να προσπαθήσει να, να καταβάλει οποιαδήποτε προσπάθεια έτσι ώστε να καλύψει αυτές τις προϋποθέσεις και αυτό είναι για το καλό και της χώρας αλλά και γενικότερα της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης εισηγητές, ο κύριος Γέλαμα από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον συνάδελφο Ιβο Βάγκελ. Πρόκειται για μια ισορροπημένη και επικοδομητική έκθεση, παρότι αναφέρει και πολλά επικριτικά ε, στοιχεία. Ε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη. Πρόκειται για ένα περιφερειακό σκηνικό το οποίο είναι ρευστό και ένα ειδικότερο σκηνικό στην ίδια τη χώρα, το οποίο διαρκώς αλλάζει είναι ιδιαίτερο ε, ρευστό. Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές ε, ότι το, εάν θέλουν ε, ε, πραγματικά στην χώρα να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει όλες οι πολιτικές ε, δυνάμεις να συμφωνήσουν, να βρουν κάποιον συμβιβασμό κυρίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις αλλά σε μια πρώτη φάση για τον σχηματισμό κυβέρνησης έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι προεντεξιακές διαπραγματεύσεις δηλαδή να ξεκινήσουν επισήμως αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, και αυτό θα γίνει ε, μονάχα ότι ε, ζητήματα με γείτονε τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτή την φάση δεν θα επηρεάσουν την διαδικασία. Μέχρι τώρα η κατάσταση στην χώρα έχει προκαλέσει κούραση και είναι γενικώ αποκαρδιωτική. Γενικώ η οι δεν σημαίνουν ε, κάτι από μόνες τους. Ε, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια εθνικής συμφιλίωσης ε, και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει ώστε όλες οι δυνάμεις να προσυπογράψουν τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βάγκελ, τον εισηγητή αυτής της έκθεσης, για το γεγονός ότι κατέθεσε όλα τα βασικά στοιχεία και ε, ανέφερε με απόλυτη σαφήνεια ότι η χώρα αυτή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Οι βουλευτικές εκλογές έλαβαν χώρα στις 11 Δεκεμβρίου. Η κατάσταση έκτοτε είναι αρκετά σταθερή. Βεβαίως ε, με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και των βουλευτών που συνέβαλαν στον εφαρμοστή Συμφωνία Πρίτσιν. Υπήρξαν πολλές προσδοκίες από τις εκλογές, γιατί οι άνθρωποι τα τελευταία δύο χρόνια ζούσαν σε μια αφύσικη κατάσταση. Άρα δηλαδή τώρα πλέον επίγουν οι μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί και η συμμετοχή των τακτικών δικαστηρίων σε έρευνες που διεξάγονται για την ελευθεροτυπία, για τη διαφθορά, για το οργανωμένο έγκλημα. Τέλος πάντων έχουν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατάσταση κατεύθυνση. Ε, βεβαίως οι διεθνωτικέ σχέσει παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. η συγητή αναφέρεται και στην πολιτική επί του προσφυγικού από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανεργία κυρίω ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκε. Ελπίζω η κατάσταση μετά τις ε, εκλογές θα συνεχιστεί πιο ομαλή χωρί να υπάρχουν ε, διακριτικέ μεταχειρήσει. Ε, προχτές ε, υπήρξε κάποια αποτυχία, αλλά εν πάση θέλω να πιστεύω ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ, Επόμενο. ο ε, εκ μέρου ε, τη ΓΚΟΕ, η κυρία Σακοράφα. Κυρία Σακοράφα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η πολιτική της επιβράβευσης όλων αυτών των αρνητικών που συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση της χώρας και που αναφέρονται πολλά από αυτά στο προσχέδιο και που ανέφερε και ο ίδιος ο εισηγητής σήμερα ο κύριος Βάγκη, από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή μόνο ανασταλτικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όσον αφορά την πρόοδο και την ευημερία του λαού του Ισφύρου. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η Φύρομ βιώνει τη χειρότερη πολιτική κρίση από το 1, το 2001 τόσο η διακοπή του πολιτικού διαλόγου, όσο και οι δυσκολίε στην εξέβρεση συνενετική λύση ώστε να ξεπεραστεί η κρίση με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναβολή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του περασμένου χρόνου, αλλά και την μέχρι τώρα αποτυχία να σχηματίσουν η κυβέρνηση, ανέδειξαν για άλλη μια φορά τη δικαχαστική πολιτική κουλτούρα και την έλλειψη συμβασμού που υπάρχει στη χώρα. Η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα υπάρχει σαφή έλλειψη πολιτικής βούλησης για να παταχθεί, ενώ όσοι νόμοι υπάρχουν δεν εφαρμόζονται, η επιλεκτική δικαιοσύνη και η ατιμορρησία όσων εμπλέκονται σε υψηλού επίπεδου υποθέσει διαφθοράς τείνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο, οι πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη στους τομείς της δημόσιας διοίκησης αλλά και των μέσων μαζική ενημέρωση συνθέτουν μια ολιστική εικόνα ανομίας, αλλά και παραπέρα οπισθοδρόμησης στα πολιτικά κριτήρια της Χάγης, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, κύριοι συνάδελφοι. Τη διαφωνία μου για το ονοματολογικό σα την έχω εκφράσει σε όλου του τόνου. Πιστεύω, κύριε Βάγκλο, ότι κάνετε μεγάλο λάθο παίρνοντα για μια ακόμη φορά θέση, αγνώντα την ιδιαιτερότητα που θα έπρεπε να επιδείξει το Κοινοβούλιο σε αυτό το διεθνέ ανοιχτό ζήτημα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η στάση αυτή, το έχω ξαναπεί, δεν βοηθάει, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να συντηρεί την άσχημη κατάσταση τη χώρα, να επιτρέπει στην πολιτική ελίτ τη Φύρομ να καλλιεργεί το έλλειμμα ανάπτυξη απαραίτητη πολιτική κουλτούρα, του σεβασμού των κανόνων δικαίου και του σεβασμού, να επενδύει στον εθνικισμό, να αντιστρατεύεται τι θεμελιώδει αρχέ τη διεθνού ένωμη τάξη και να αγνοεί την έλλειψη πρόοδου στη σχέση καλή γειτονία. Τελικά, κατά την άποψή μου, το θέμα, κύριε είναι να θέλει και ίδια η Φύρομ να προοδεύσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας. Okay, we go into the Greens, Mr. Ε, πάμε τώρα στους πράσινους, ο κύριος Μαζαρίτσε. Ε, αλλάζω πάλι ιδιότητα. Τώρα είμαι σκιώδη ηγητή ε, για το θέμα που συζητάμε και να ευχαριστώ τον Στάφο κύριο Βάγκελ ε, για την πολύ επαγγελματική και ισορροπημένη έκθεση. Ε, εγώ συμφωνώ, πολύ λίγα θέλω να σχολιάσω. Το ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς πιστεύουμε, όπως λέει και το κείμενο, ότι οι διμερείς διαφωνίες δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Εντάξει, υπάρχουν άλλα εμπόδια, αλλά ας μην είναι και αυτό άλλο ένα, οι διμερείς διενέξεις. Ε, θεωρούμε ότι ε, θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, αυτό το θέμα το διμερέ να λυθεί από ένα διεθνέ δικαστήριο. Εμεί αυτό πιστεύουμε. Στην ΦΥΡΟΜ υπάρχει διαφθορά και ε, οργανωμένο έγκλημα, όπως και σε άλλες χώρες των Δυτικών, Δυτικών Βαλκανίων. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζονται στην ίδια τη χώρα και ε, θεωρώ ότι επ' αυτού ίσως υπάρχουν κάποιες ελπίδες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω τις ε, συστάσεις της μόνιμης επιτροπής της Βέρνης, ε, ένα σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα ε, στα Βαλκάνια εφίσταται, είναι θέμα η προστασία του περιβάλλοντος. Η μόνιμη αυτή επιτροπή καλεί τη μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος μέχρι να υπάρξει ε, μια στρατηγική χάραξη, μια στρατηγική επί Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα καταθέσουμε σχετικές ε, τροπολογίε. Και έχουμε τώρα πέντε ομιλητές, ε, ένας από κάθε ομάδα. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την εργασία του συναδέλφου Ιβο Βάγγελ. Έθεσε την προσοχή τους στα σημαντικότερα θέματα ε, όντως. Αυτή τη στιγμή στην χώρα αυτή η βαθιά πολιτική κρίση δυναμητίζει τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα. Ε, ο διπολισμός, η πόλωση του πολιτικού ε, σκηνικού ε, δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, δείχνουν ότι οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει μπλοκαριστεί και επομένως δεν προχωράει καμία μεταρρύθμιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναέρθουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να βρεθεί μια κυβέρνηση έτσι ώστε να αρχίσουν να δουλεύουν σοβαρά ε, με τρόπο ώστε ε, η φύρομαι να ξαναμπεί στην ευρωπαϊκή τροχιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ε, σημαντικό και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να μεταδώσει τούτη η έκθεση. Ο κύριος Φλέκενστάιν, του τους δημοκράτε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Βάγκελ για την έκθεσή του. Μόνο επιτρέψτε μου να πω κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Διότι κυκλοφορούν φήμε στη Μακεδονία ότι σε αυτό το κοινοβούλιο και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν του είναι σημαντικό το ποιος κυβερνάει όσο υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία. Κατά πόσον ε, κυβερνούν οι συντηρητικοί με τους αλβανόφωνους ή οι σοσιαλιστές με τους αλβανόφωνους. Σημασία έχει, αυτό που σε ενδιαφέρει, είναι να έχουν μια σταθερή κυβέρνηση η οποία θα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο, την ευρωπαϊκή πορεία. Και οι μεταρρυθμίσεις, όπως συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία του Πρίτσινο, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και η πολιτική αυτού του ειδικού εισαγγελέα. Αυτό παίζει ρόλο. Αν δηλαδή θέλει κανείς να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Το θέμα δεν είναι να πούμε είμαστε υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όταν δύο πλευρέ δείχνουν την ίδια σταθερότητα αν ο ένα θέλει να έρθει στην Ευρώπη. Ο κ. Παπαδάκης παρακαλώ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ε, οι δηλώσει του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου κ. Ταγιάννη σε προηγούμενη επίσκεψή του στη χώρα αποδείχθηκε πω είναι συνδεδεμένε με άλλε ανησυχητικέ ενέργειε. Για παράδειγμα η έκθεση προόδου παραβλέπει προκλητικά και επανειλημμένα την επίσημη ονομασία τη χώρα πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργούν και ταυτόχρονα στηρίζουν δυνάμει που προωθούν αλυτρωτισμού, αμφισβητήσει κυριαρχικών δικαιωμάτων, εθνοθρησκευτικού διαχωρισμού. Οι δε εκκλήσει για πιο ενεργό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με εμπλοκή τη ΥΠΑ εκπροσώπου έχουν στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου σε ανταγωνισμό με ρώσικα συμφέροντα στα Βαλκάνια. Εργαλείο σε αυτή την υπόθεση αποτελεί και η εν λόγω έκθεση και νέα αντεργατικά μέτρα προτείνει η έκθεση και για τον λαό τη ε, πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Η έκθεση επίση βαφτίζει επικοδομητική συνεργασία τη Πούγου Δουμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό, ομολογώντα ότι συνεργάστηκαν για το απαράδεκτο κλείσιμο των συνόρων με άγρια καταστολή στου πρόσφυγε οι οποίοι εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Οι λαοί τη περιοχή κόντρα στον εθνικισμό, τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου και τα εμπεριστικά σχέδια να παλέψουν για τα δικά του συμφέροντα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια και το σύστημά του. Ευχαριστώ. Mr. for one minute. για Ρίσεις. Στην έκθεση στο σημείο Α, σελίδα 4, αναφέρεται Parliamentary elections held in Macedonia had a very high turnout. Στο σημείο 17, στη σελίδα 6, αναφέρεται πάλι risk to the Macedonian economy. Και στο σημείο 22, σελίδα 7, welcome Macedonians uh, international cooperation and things like this. Ε, θέλω επίσης και εγώ να αναφερθώ στην ε, δήλωση του κ. Ταγιάννη, αλλά της περασμένης Τετάρτης, ο οποίος αναφέρει ότι η πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι το σώμα αναγνωρίζει εισαγωγικά, διαβάζω όπως το έγραψε, ως μόνη ονομασία της χώρας διεθνώς αναγνωρισμένης ως πρώην, δημοκρατι... ως Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Φύρομ. Και θέλω να πω, ε, η έκθεση ενώ ενώ στον τίτλο της έχει report για το former, former Yugoslavian Republic of Macedonia γιατί αναφέρεται σε Μακεδονία μέσα στο κείμενο. Το δεύτερον, στο σημείο F της σελίδα 4 μιλάει για bilateral disputes uh, should not, should not uh, uh, represent uh, an obstacle in the opening of the accession negotiations. Θέλω να θυμίσω στον κύριο ε, εισηγητή Κλίνο ότι είναι διεθνές θέμα, δεν είναι διμερές θέμα και αυτό αναφέρεται στο ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το οποίο πρέπει να δει είναι το Resolution 817 του 1993 και 845 του 1993 και παρακαλώ πολύ τον κύριο εισηγητή να τα διορθώσει. We go to Mr. Ο κύριος Επιτήδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω και εγώ στην έκθεση το σημείο εκείνο το οποίο αναφέρεται στις ε, διμερείς ε, διαφορές και ότι αυτές δεν πρέπει να ε, αποτελούν εμπόδιο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δύο σημεία εδώ. Το ένα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, μόνο η διαφορά των Σκοπίων με την Ελλάδα για το θέμα του ονόματος. Και το πιο σοβαρό είναι αυτό το οποίο ήδη αναφέρθηκε ότι το θέμα δεν είναι διμερές, είναι διεθνές. Τα Σκόπια έχουν υποχρέωση σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής, του, της Γενικής του ΙΕ σε όλες τις δραστηριότητες τους να εμφανίζονται ως πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εφόσον κάνουν αυτή την παραβίαση, από εκεί και πέρα είναι αυτές υπεύθυνοι για το ότι υπάρχει ε, παρεμπόδιση της, ε, της ανάξεως των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και από το σημείο αυτό επίσης θα ήθελα να καταδικάσω την ε, ε ατυχή ε, ε, ε, έμπνευση που είχε ο κύριος Σταγιάννη να ονομάσει τα Σκόπια Μακεδονία δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα άλοθη στη γειτονική χώρα να μην σημειώσει πραγματική πρόοδο. Ευχαριστώ. Then last uh, Κυρία Τσουίκα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάγκλ για την ε, δέσμευσή του και την προσπάθεια που κατέβαλε για την έκθεσή του, αλλά επίσης και σε όλο το διάστημα που εργάστηκε για να μπορέσουμε να επιληθεί τα προβλήματα αυτά σε σχέση με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία. Ήταν πολύ επαγγελματική η εργασία του και όπως είπε και ο κύριος Φλέγκενστάιν, είναι σωστό ότι οποιαδήποτε και να είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει την σταθερότητα της χώρας αυτής, ώστε η πρώην Δημοκρατία να επανέλθει στον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να παίξει και ρόλο στην περιφερειακή συνεργασία που είναι απαραίτητη για την πορεία προς την Ευρώπη. Θα πρέπει να επιληθούν όλες οι διμερείς διενέξεις με έναν τρόπο ικανοποιητικό και τα εκρεμή ακόμα θέματα με την Βουλγαρία και αυτά θα πρέπει να επιληθούν σε διμερές επίπεδο. Χρειάζεται να υπάρξει μια σταθερότηση και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει συμφωνία, να τηρηθεί συμφωνία του Πρεζίνο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 ε, αυτό το θέμα της ε, ε, Μακεδονίας είναι γνωστό. Η Ελλάδα έχει βέτο όσον αφορά τα θέματα αυτά και φαίνεται ότι από όλες τι πολιτικές ομάδες όλοι έχουν την ίδια άποψη. Είναι on block. Τι να σας πω, εδώ μιλάμε για Μακεδονία, έτσι είναι και μην προσπαθείτε να μας πείσετε Κοιτάξτε και στα νέα μας και στις εφημερίδες μας εμείς πάντα μιλάμε για τη Μακεδονία. Καταγράψτε το, ε, σημειώστε το. Ε, εντάξει έχετε ε, δικαίωμα βέτο, το ασκείτε πάρα πολύ ωραία, αλλά τα πράγματα έτσι είναι. Πέρασε και ο αιώνας και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Λυπάμαι, λυπάμαι γιατί νομίζω ότι το θέμα μας θα έπρεπε να είναι ο λαός της Μακεδονίας και όχι κάποια θέματα τα οποία άπτονται της ιστορίας και μάλλον της μυθολογίας. Κομισιόν θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Βοβάγγελ για αυτήν την ε, έκθεση. Ε, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό να στείλουμε ε, σωστά μηνύματα στην χώρα. Θεωρούμε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει σωστά τα ευρήματα της έκθεσης για τη χώρα του 2016. Εμείς σχετικά με την πολιτική κατάσταση, έχουμε εκφράσει την, ε, ε, τον προβληματισμό μας, έχουμε εκφράσει τον προβληματισμό επίσης ε, για την κακή λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Ο κύριος Βάγκερ, ο κύριος Κούκαν και ο κύριος και ο κύριος Φλέκενστάιν σωστά έχουν τοποθετηθεί όσον αφορά τα θέματα αυτά. Οι πρόορες εκλογές ήταν μέρος της συνολικής συμφωνίας αλλά αποτέλεσαν μόνο την αρχή. Τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε <laughs> να σχηματιστεί μια ε, σταθερή κυβέρνηση. Θα πρέπει η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση να συνεργαστούν αγαστά έτσι ώστε ε, να ε, μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα και η χρονική υστέρηση και η Θα πρέπει οπωσδήποτε εμείς να δούμε τις ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, θα πρέπει να δούμε επίσης ότι το γραφείο της ε, εισαγγελία δίνει τους πόρους και τις, θέτει τις προϋπο, του, του ειδικού εισαγγελέα και θέτει και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ε, ειδικές προτάσεις της ε, Κομισιόν. Εμείς ε, είμαστε σαφείς όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε η χώρα να ξαναμπεί σε ευρωπαϊκή τροχιά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε την επιτήρηση της κατάστασης, να βοηθήσουμε την χώρα και να υπάρξουν τακτικές ενημερώσεις του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητή θέλει μήπω να ξαναπάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Κύριος Βάγκλ, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τα σχόλιά τους σε σχέση με την εκθεσή μου. Εγώ θέλω να σας εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου για όλες τις τροπολογίες που καταθέσατε. Θέλω να πω όμως και το εξή ακόμα, στο περιθώριο της συζήτηση για το όνομα της χώρας αυτής. Εάν πρόκειται για διεθνές θέμα, παγκόσμιο θέμα ή διμερές θέμα ανεξάρτητα από τη φύση του θέματος αυτού, νομίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε ακόμα αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιληθεί το ταχύτερο δυνατό και χρειάζεται μια πιο έντονη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιληθεί το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα αυτό μόνο στα Ενωμένα Έθνη. Τα Ενωμένα Έθνη είναι μακριά μας, αλλά η χώρα αυτή είναι πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αν εμποδίσουμε λοιπόν να υπάρξει η προσέγγιση της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσουμε και ένα υψηλό τίμημα. Κατανοώ βέβαια τη θέση των Ελλήνων συναδέλφων, οι οποίοι έχουν εκφράσει με σαφή τρόπο και κοινοβουλευτικό τρόπο τις αντιρρήσεις τους. Καταλαβαίνω τις απόψεις που έχουν διατυπώσει αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η πλειοψηφία των βουλευτών που βρισκόμαστε εδώ και που εκπροσωπούμε τις χώρες μας θεωρούμε ότι η χώρα αυτή που βρίσκεται στα Βαλκάνια ονομάζεται Μακεδονία. Αυτό είναι η δική μας εικόνα της πραγματικότητας ότι η χώρα αυτή λέγεται Μακεδονία. στις 28 ε, Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε, 12 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Περνάμε τώρα στην έκθεση για το Μαυροβούνιο και δίνω για 3,5 λεπτά το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Τένοκ. Είναι η πρώτη εξέταση του θέματος, οπότε θα έπρεπε να έχω 5 λεπτά. 5 χρόνια από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 26 από τα 33 κεφάλαια έχουν ανοίξει, 3 έχουν κλείσει προ... προσωρινά. Υπήρξε μεγάλη πρόοδος στη χώρα αυτή και είναι σαφής ο δρόμος που ακολουθεί προς την ένταξη και πολύ θετική η πρόοδος. Κεφάλαιο κεφάλαια 23 και 24 για τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών είναι σαφής η πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί και οι μεταρρυθμίσεις μετά από την περσινή μου έκθεση που ήταν πολύ σημαντική. Έλαβαν χώρα κοινοβουλευτικέ εκλογέ στο Μαυροβούνιο, άλλαξε πρωθυπουργό, συνάντησε τον κύριο Μπράγκοβιτ την προηγούμενη εβδομάδα και υπεγράφει ένα πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έγιναν εκλογέ με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με καταγραφή όλων των ε, ψηφοφόρων και ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησή του, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι καλύτερο από το σύστημα που τουλάχιστον δική μου χώρα έχει. Δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση λοιπόν μετά τις εκλογές που επέτρεψε σε πρώην εκπροσώπους αντιπολίτευσης να λάβουν σημαντικά και κέρια υπουργεία και έτσι με τον τρόπο αυτό υπήρξε και κάποια εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει υπερβολική εξουσία του κυβερνώντος κόμματος οι διεθνεί παρατηρητέ είπαν ότι ήταν αδιάβλητε και δίκαιε οι εκλογέ και υπήρξε σεβασμό των βασικών ελευθεριών. Υπήρξε κάποια ανησυχία για το γεγονό ότι ε, έκλεισαν ορισμένα κοινωνικά μέτρα διαδικτύωση στη μέρα των εκλογών, αλλά αυτό δεν είχε μεγάλη επιρροή στι εκλογέ. Εξακολουθούν οι έρευνε στα θέματα αυτά, αλλά υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ κυβερνητικών και αντιπολιτευτικών κύκλων ότι οι επιθέσεις οι οποίες έλεγαν κατά του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσουκάροβιτς ήταν μια πραγματική απειλή. Εγώ εξακολουθώ να ανησυχώ για την κατάσταση λοιπόν που επικρατεί στη χώρα αυτή που καταδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που προσπαθεί να ασκήσει η Ρωσία στο Μαυροβούνιο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι σαφές ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια ιδίως από τη Ρωσία να εμποδίσει την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ και να εμποδίσει το δρόμο του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο όλα τα πολιτικά κόμματα να αγωνιστούν μέσα σε μια καθαρή δημοκρατική διαδικασία στο κοινοβούλιο του. Η συνέχιση του μποϊκαταρίσματος του Κοινοβουλίου από την αντιπολίτευση είναι κάτι το οποίο απογοητεύει και υποσκάπτει την αξιοπιστία της δημοκρατικής διαδικασίας του Μαυροβουνίου. Όπως πάντα, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε μια καλή ισορροπία στην έκθεση της Επιτροπής μας ώστε όλες οι πολιτικές ομάδες να μπορέσουν να προσυπογράψουν αυτήν την ε, έκθεση όπως και τα προηγούμενα χρόνια και είναι η 7η χρονιά που είμαι μόνιμος εισηγητής. Πάντα είχαμε καταφέρει να αποσπάσουμε μια μεγάλη και ευρεία συνένεση. Το Μαυροβούνιο πάντα είναι μια, ένα θετικό παράδειγμα και μια χώρα η οποία αντίθετα από τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα Εφόσον και το Μαυροβούνιο θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εφέτο, θα πρέπει εμεί να υποστηρίξουμε αυτή την αίτηση του Μαυροβουνίου. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο διαφορετικά ε, όργανα, αλλά ουσιαστικά δείχνουν και τις κοινέ αξίες και την ευρωατλαντική σύνδεση των χωρών μας. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτήν την, ε, αυτό το θεματολόγιο και ενώπιον της αλλαγής ε, κυβέρνησης στις ΗΠΑ Ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι θα δεχθούν το γεγονός ότι θέτω τον ΝΑΤΟ στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τις απόψεις των άλλων σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ. On behalf of Mrs. Η ε, κυρία Μάγερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα μιλήσω εξ ονόματο ε, τη Αναλύης Νατότς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Τσάρλ Τόνοκ ε, για την ε, καλή συνεργασία στη διάρκεια των συναντήσεων των σκιωδών εισηγητών. Στην έκθεση αναφέρονται σημαντικά συζητήματα, κυρίω όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την παρατήρηση, την έκθεση των εκλογών από πλευρά τη υπηρεσία υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Ε, ε, λαμβάνουμε υπόψη μα όλα τα σημεία τα οποία αναφέρει αυτά. Ε, αυτή η έκθεση θα πρέπει να βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση, κυρίως δε ε, ανησυχητικό είναι το μπλοκάρισμα αυτό τη αντιπολίτευση. θα πρέπει ε, οπωσδήποτε και είναι θεμελιώδου σημασία να υπάρξει πλήρη διαλεύκανση ε, της ε, πράξη ε, Επίση, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ε, το μεγαλύτερο ποσοστό των Μαυροβουνίων επιθυμούν ε, την προσέγγιση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό το ΕΛΚΑ. Ε, η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του κυρίου Κόβατς θα πω ότι ε, συγχαίρουμε τον κύριο Τάνοκ για την εργασία του. Όντως το Μαυροβούνιο ε, αποτελεί, ε, είναι μια χώρα η οποία έχει δώσει καλά αποτελέσματα στην περιοχή των Βαλκανίων. Δυστυχώς ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων δεν έχει ληφθεί υπόψη στην έκθεση εδώ. Είναι γεγονός ότι η χώρα έχει αντιμετωπίσει κάποια ε, προβλήματα. Ο κύριος Κόβατσεκ αναφέρεται σε οικονομικά προβλήματα, αναφέρεται σε προβλήματα του δικαστικού ε, ε, συστήματος, προβλήματα που συνδέονται με την ανεργία, επίσης θέματα τα οποία σχετίζονται με την κυκλοφορία κεφαλαίων. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει κάποια τμήματα νομοθεσίας να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα, καθώς επίσης και να υπάρξουν και κάποιες τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις. Είναι ε, γεγονός ότι κυρίως το δικαστικό σύστημα θα πρέπει να προοδεύσει η καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, του οργανωμένου εγκλήματος και της ε, εγκληματικότητας και άλλα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σκιώδης ηγητής κύριος Κόβατσεκ ε, συγχαίρει την ε, χώρα ε, όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική και την ευθυγράμμιση με τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την εξωτερική πολιτική και επίσης η αρμόδια αρχή του Κοινοβουλίου έχει... Συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Αντρουλάκη που δεν βρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση. Το Μαυροβούνιο παραμένει ο πρωταθλητής στο Δυτικό Βαλκανίο. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες χώρες και η δυναμική αυτή πρέπει να διατηρηθεί. Δυστυχώ όμω, γεγονότα όπως η αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση την ημέρα των εκλογών και η απόφαση μέρους της αντιπολίτευσης να απέχει από τις εργασίες του Κοινοβουλίου προκαλούν ανησυχία. Θα ήταν άδικο μια ενδεχόμενη περίοδος πολιτική αστάθεια να ακυρώσει τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει. Είναι ανάγκη να υπάρξει άμεση διαλεύκαση της αποτυχεμένης τρομοκρατικής επίθεσης. Είναι απαραίτητο επίσης η αντιπολίτευση να συμμετάσχει κανονικά στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Παρά τις όποιες δυσκολίες έχουν παρουσιαστεί η ενταξιακή πορεία της χώρας έχει μείνει σχετικά ανεπηρέαστη. Χαρακτηριστικά πρέπει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα εργασιών της που υιοθετήθηκε την Παρασκευή οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο παραμένουν πρώτη προτεραιότητα. Επιπλέον, το άνοιγμα του κεφαλαίου 19 σχετικά με την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση μπορεί να δώσει το πλαίσιο για περαιτέρω προσπάθειε μείωση τη ανεργία και ιδιαίτερα τη ανεργία των νέων. Στο θέμα του ΝΑΤΟ, απλά θα ήθελα να αναφέρω πως αν και είναι σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, η είσοδος της στη Συμμαχία, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία και δεν πρέπει να συγχαίεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ, για το πολύ καλό σχέδιο ψηφίσματος που έχει προετοιμάσει, θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες σχετικά με τα θέματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. On behalf of the group, Mr. Ο κ. Βάντος, Ράντος από την ομάδα του ALDE. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την θαυμάσια έκθεσή του και την πολύ καλή συνεργασία που είχε με όλους μας στο Μαυροβούνιο είναι η χώρα η οποία είναι πιο έτοιμη για την ένταξη της Ευρω... προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει και προβλήματα, ιδίως στρατηγικού χαρακτήρα προβλήματα. Υπάρχει το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η διαφθορά, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Η εκλογική διαδικασία είχε επίσης προβλήματα, παρά το γεγονός ότι τελικά όλα πήγανε καλά. Είναι μια χώρα που βρίσκεται ακόμα σε δημοκρατική πορεία. κάτι ακόμα που είναι σημαντικό. Η ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί και η οποία εμποδίζει τη σωστή λειτουργία αυτής της χώρας. Θα ήθελα να αναφερθώ στην επίθεση αυτή που έγινε κατά των θεσμών του Μαυροβουνίου που έλαβε χώρα την ημέρα των εκλογών θα μπορούσε να είχε τραγικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις, σε εξεγέρσεις, σε μια βαθιά κρίση. Εξακολουθεί όμως η δυνατότητα μιας αντιπαράθεσης γιατί συνεχίζεται το μποϊκοτάρισμα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και υπάρχουν και ξένες αναμίξεις. Πρέπει οι έρευνες λοιπόν να γίνουν με σωστό τρόπο για να ξέρουμε ποια ήταν η μαύρη χείρ η οποία δημιούργησε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Δεν έχουμε κάποιον άλλο μιλτή Α, όχι, συγγνώμη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ αντικαθιστώ την κυρία Λούνατσεκ, η οποία δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την πολύ καλή του έκθεση για το Μαυροβούνιο και θέλω να προσθέσω και κάποια δικά μου σημεία σε αυτό. Εμείς σίγουρα συμμεριζόμαστε αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής σε σχέση με την ε, επίθεση που έγινε. Πιστεύουμε επίση ότι η Ρωσία προσπαθεί να αναμειχθεί και να επηρεάσει τα πράγματα στο Μαυροβούνιο και αυτό είναι ανησυχητικό. Κάτι επίση ανησυχητικό, όσο και η επίθεση είναι το γεγονό ότι μπλοκαρίστηκαν τα κοινωνικά μέσα διαδικτύωση την ημέρα των εκλογών. Κάτι φυσιολογικό σε χώρε όπω η Κίνα ή η Ρωσία, αλλά όχι σε μια χώρα που είναι υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαλάβει κατά την άποψή μου και η έκθεση. Για αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5, ιδίω στην ε, καταγραφή συνομιλιών, υπάρχουν και άλλε περιπτώσει ε, υποκλοπή τηλεπικοινωνιών που μέχρι σήμερα δεν έχουν διαλευκανθεί αυτές οι υποθέσεις υψηλού προφίλ και που εμπλέκουν ε, πολιτικούς και από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ίσως τέλος για το περιβάλλον θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ καλό του κείμενο. Θα πρέπει με σαφή τρόπο να αναφερόμαστε στην διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει να κάνει με το περιβάλλον για το Μαυροβούνιο και να αναφερθούμε και στα υδροελεκτρικά έργα όπως και σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι το άγριο West, το Wild West, το μαυροβούνιο για τους επενδυτές. Δεν μπορούν όμως να συνεχίσουν αυτά τα πράγματα να είναι χωρίς κανόνες. Και επίσης το φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερη προσοχής, το όμορφο φυσικό περιβάλλον του Μαυροβουνίου, να έχει ειδική προσοχή. Ο κύριος Κούκαν από το ΕΛΚ επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και με ευγνώμων στον εισηγητή για την αφοσίωση με την οποία παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο Μαυροβούνιο. <coughs> το Μαυροβούνιο πέρσι εξέλεξε μια κυβέρνηση η οποία είναι υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζει τον ευρωατλαντικό του δρόμο. Επειδή αυτό είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας, εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα αυτή την επιλογή. Πρέπει να καταγράψουμε επίση και την υποστήριξη των πολιτών για την, ε, τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαυροβουνίου, η υποστήριξη αυτής της πορείας φτάνει το 80%. Λείπαμε που η αντιπολίτευση απέχει από το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι το κοινοβουλευτικό έργο θα επαναληφθεί ώστε να μπορέσει να προωθηθεί όλο το πολιτικό θεματολόγιο. Η αντιπολίτευση πρέπει να βρίσκεται μέσα στο Κοινοβούλιο και όχι έξω από αυτό. Οι προσπάθειες λοιπόν για την ένταξη θα πρέπει να ακολουθηθούν και από την πρέπουσα μέρημνα για την εσωτερική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και, των, και της διαφθοράς και τη βελτίωση των μέσων ενημέρωσης. Το Μαυροβόνιο αποφάσισε να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και το υποστηρίζουμε και εμείς. Η αυξανόμενη όρεξη της ρωσικής αρκούδας στην περιοχή μας ανησυχεί. Αλλά εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε και όχι να αποθαρρύνουμε το Μαυροβούνιο από το να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο ε, Τάνοκ ε, σχετικά με την ε, έκθεσή του, την γνωμοδότησή του το περιεχόμενο της οποίας μας βρίσκει σύμφωνους. Ε, η πλήρη ε, εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τις ε, αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτα απαραίτητη για την, τα Δυτικά Βαλκάνια και ιδιαίτερα το Μαυροβούνιο και αυτό το είπαμε και στον κύριο Μάρκοβε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πρέπει το Μαυροβούνιο να έχει την δυνατότητα ελεύθερα να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση και την εξέλιξη και εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι όσον αφορά την πόλωση που υπάρχει εκεί. Ε, θα πρέπει ε, οπωσδήποτε οι αποφάσεις να λαμβάνουν και η αντιπολίτευση να συμμετάσχει ε, σε την πολιτική ζωή του τόπου επιστρέφοντας στο κοινοβούλιο εκεί όπου ανήκει. Θα έχει ξεκινήσει η πρόοδος και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει συνέχεια ε, ρητά ε, όσον αφορά την ε, το κράτος δικαίου θεωρούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο έτσι όπως τα αναφέρετε. Παραμένει η διαφθορά ένα κυρίαρχο μέλημά μας και μας προβληματίζει ιδιαίτερος όπως μας προβληματίζουν και εμπόδια στην λειτουργία του κράτους δικαίου. Τέλος, θα πω δύο λόγια για την οικονομία. Το Μαυροβούνιο ε, θα πρέπει ε, γρήγορα ε, να, και επιγόντως μάλλον να τροποποιήσει την φορολογική του πολιτική. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέσω επιπλέον πρόσθετων μεταρρυθμίσεων να μειώσει τις δαπάνες. Αυτά και σας ευχαριστούμε πολύ για τη θέση που έχετε πάρει όσον αφορά το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο θέλει, Κύριε Τάνοκ, θέλετε να πάρετε το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ναι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές ε, και κυρίως ε, τον φίλο Κούκαν για τα καλά λόγια και επίσης να πω ότι μαζί με την κυρία Λούνατσεκ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Μαυροβούνιο. Επίσης ε, ε, θα ήθελα ε, να αναφερθώ και σε την ευθυγράμμιση του Μαυροβουνίου όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας αντίθετα από τη γειτονική Σερβία. Είναι αλήθεια κυρία Σουίτσα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις για το μέλλον. Βλέπουμε τα θέματα αυτά, τα μελετούμε ε, σε αιτήσια βάση. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες είναι πολύ σωστέ όσον αφορά την ελευθεροτυπία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οποτεδήποτε ε, μπορώ θα τα υποστηρίξω. Ε, και βεβαίως να ευχαριστήσω και την κυρία Ντότσο για την συνεργασία της. Είναι πάρα πολύ θετική η προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 2 Φεβρουαρίου και με αυτό ολοκληρώθηκε το δημόσιο ε, τμήμα της συνεδρίασης, η οποία θα συνεχιστεί και κλεισμένο των θυρών. Ευχαριστώ πολύ.